Σας καλωσορίζω όλους. Ο πρόεδρος μας θα έρθει λίγο αργότερα κατά το δεύτερο τμήμα της συνάντησης αυτής, της σημερινής. Βρίσκεται σε μια συνάντηση με τον πρώην Επίτροπο Φίσλερ και μάλλον θα παρευρεθεί μετά τις 4. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, στο προσχέδιο. Θα ήθελα να σας πω ότι για τεχνικούς λόγους δεν, δεν μπορούμε να έχουμε διερμηνία προς και από όλες τις γλώσσες. Δεν έχουμε φινλανδικά και λιθουανικά σήμερα. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θεωρώ ότι Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν σχόλια ως προς τα πρακτικά, ε, στο τέλος της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε εγκεκριμένα τα πρακτικά της 28 29 φεβρουαριου Όπως γνωρίζετε, η συνάντησή μας, η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στην ε, έκθεση Dorfman για τα ε, αρωματισμένα αμπελοϊνικά προϊόντα και όπως ξέρετε μαζί με την Envy συμμετέχουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση, δυνάμει του άρθρου 50. Υποβλήθηκαν 24 τροπολογίες στη γνωμοδότηση αυτή, στο προσχέδιο γνωμοδότησης. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντόρφμαν, τον εισηγητή μας. Χέρμπερτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε την ε, ψηφοφορία. Θα ήθελα μόνο να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω θερμά τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για αυτό το τόσο τεχνικής φύσεως θέμα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Πρόκειται λοιπόν για την ε, επεξεργασία των υφιστάμενων οδηγιών ε, σχετικά με την προέλευση των ε, αρωματικών, αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τομέα που μιλάμε για περίπου εκατομμύρια στρέμματα παραγωγής, ε, κυρίως στη Μεσόγειο. Για άλλη μια φορά λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και νομίζω ότι τώρα πλέον έχουμε μια ε, πολύ καλή πρόταση και ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί επίσης. Ας προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρήσουμε τώρα στις ε, ψηφοφορίες. Μπορεί να χρειαστεί να... μερικές να τι ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ο κ. Καπολασάντος θέλει να πάρει το λόγο. não, tenho o meu cartão de voto no meio de, de algumas centenas deles e pedi-lhe que considerasse um voto. Δεν ε, έχω μαζί μου την κάρτα, γι' αυτό να συμπεριλάβατε και τη δική μου ψήφο, δηλαδή μία επιπρόσθετη ψήφο από τους σοσιαλιστές. Μάλιστα. Ε, θα προσπαθήσουμε χωρίς ηλεκτρονικά μέσα να ψηφίσουμε. Μπορώ να του δώσω την κάρτα μου αν θέλει ο κύριος Κάπουλας αντός; Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Μόνο σαν πιστοτική κάρτα είναι η κάρτα ψηφοφορίας. Εγώ έχω τρεις, αλλά μπορώ μία να χρησιμοποιήσω. Οπότε, ας περάσουμε στη ψηφοφορία. Και Σιλβέστρη. Εγώ θα ήθελα και εγώ να του δώσω την ε, κάρτα μου, αν μου δώσει μια πιστοτική που έχει στο πορτοφόλι του. Πολύ ευχαρίστως θα άλλαζα την κάρτα μου με μια πιστοτική, την κάρτα ψήφου. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Έχει έρθει και η άνοιξη, αλλά ας περάσουμε στη ψηφοφορία. Τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Σιλβέστρης υπέρ. Ταυτόσημε με την 25. Τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Λοιπόν, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 έχει αποσυρθεί. Οπότε την 26 ψηφίζουμε. Πάλι από, το, από την κυρία Σιλβέστρη. Υπέρ. Τις 27. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σχεδόν ομοφόνος. Τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 του εισηγητή. Και υπάρχει και μια προφορική τροπολογία. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος στην αρχική μου έκθεση. Το 7, το οποίο περιλαμβάνεται τώρα στην αρχική πρόταση ήταν 7%, ε, παλαιότερα ήταν 7,5%. Πρόκειται για τεχνική προσαρμογή έτσι ώστε να υπάρχει ε, εναρμόνιση των, ε, της περιεκτικότητας των αρωματικών, των αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων. Είναι τεχνικής φύσεως η αλλαγή αυτή. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση. Ποιο είναι λοιπόν υπέρ τη τροπολογία αυτή μαζί με την προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Σιλβέστρη. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε, είναι ταυτόσημη. Η 6 έχει, απο, έχει αποσυρθεί. Και για την 7 το ίδιο ισχύει. Τροπολογία 8 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. 30. Τροπολογία 30. Λαβία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Του εισηγητή. Υπέρ. Υπέρ της 10 λοιπόν. Κατά. Άλλη μια φορά λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη. Υπέρ της τροπολογίας 10. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 έχει αποσυρθεί. 34 υπέρ. Υπέρ λοιπόν της 34, Λαβία. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Τροπολογία 11. Του εισηγητή. Υπέρ. Είναι ταυτόσιμη με την 35. Υπέρ λοιπόν της 11. Άλλη μια φορά ζητά συγγνώμη ο Πρόεδρος γιατί υπάρχει σύγχυση. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικός. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας. Κύριε Καπούλα Σάντο, ψηφίσατε. Κατά. Ωραία. Εντάξει. Οπότε απορρίπτεται. Απορρίπτεται η τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στην... Τροπολογία 32. Ράμερς Λάιον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 Λαβία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Τομασεύσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Δεν θα την ψηφίσουμε. Πάμε στη 13 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Μία ακόμη φορά, λοιπόν, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία 13. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Απορρίπτεται. 19-17. Κύριε Καπούλα Σάντος, καταψηφίσατε. 37 έχει αποσυρθεί. 38. Υπέρ της 38. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 Τομασεύσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40 στο Γιάννο. Υπέρ. Τη τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 του εισηγητή και πάλι. Υπέρ της τροπολογίας 15. Κάτα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 18. Και πάλι του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με πλειοψηφία. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Συγγνώμη. Ή δεν βλέπω καλά ή δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Εγκρίνεται, εν πάση περιπτώσει. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στα εκτιμώντας. 5. Τροπολογία 21 δηλαδή, το Μασεύσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22, το Μασεύσκι και πάλι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23, το Μασεύσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότηση όπω τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά. Νομίζω τελειώσαμε να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. proszę Państwa, szukam tych swoich notatek. Βλέπω τις σημειώσεις μου, αγαπητοί συνάδελφοι, για να βρω το σωστή σελίδα. Yes. Yes. Να περάσουμε λοιπόν στο εργαστήριό μας που αφορά τα προβλήματα αστάθειας της αγοράς. Εργαστήριο για την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς, μηχανισμοί ΚΟΑ και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Zapewne nasza dyskusja przyczyni się do Νομίζω ότι έτσι θα εμπλουτίσουμε τη γνώση μας και την κατανόηση της ε, αναθεώρησης ε, της μεταρρύθμισης κοινής γεωργικής πολιτικής, ειδικότερα ε, αναφέρομαι στην έκθεση Κάπουλα Σάντος και Ντοντά για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον εμπειρογνώμονά μας, τον Αλεξάνδρο Γκοέν, από το ε, Γαλλικό Ινστιτούτο ε, Γεωργικής Έρευνας που μας παρουσιάσει τις απόψεις του για αυτό το ε, θέμα που εξετάζουμε όσον αφορά δηλαδή τη ρύθμιση των μηχανισμών ΚΟΑ και είμαι βέβαιος ότι θα απαντήσει στα σχόλια και τις ερωτήσεις μας κατόπιν της παρουσίασής του. Θα ήθελα όμως να του δώσω το λόγο. Κύριε Γκουάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας καλημερίζω όλους. Θα σας παρουσιάσω τη μελέτη μου για την αστάθεια των γεωργικών αγορών και την ανάλυση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα ε, ΚΑΠ 14-20, Υπάρχει γραπτή έκθεση, δηλαδή σε μια πρώτη φάση θα ήθελα να σας υπενθυμίζω γιατί χρειάζεται δημόσια δράση σε αυτό το τομέα. Καταρτίστηκαν πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την αύξηση τιμών και την αστάθεια των γεωργικών τιμών παγκοσμίω. Παγκοσμίως. Και υπήρξαν προβλέψεις που διαφέρουν οι μεν από τις ε, δε. Δηλαδή κανείς πάντα μπορεί να αιτιολογήσει ένα μέτρο το οποίο προτείνει. Εγώ προσπαθώ να πλαισιώσω συνεκτικά αυτό το τομέα, γι' αυτό υπενθυμίζω αυτά που έχει αναγνωρίσει ο οικονομικός τομέας γιατί δηλαδή χρειάζεται δημόσια παρέμβαση. Σε μια δεύτερη φάση θα συγκρίνω αυτά τα οικονομικά επιχειρήματα, τον οικονομικό κλάδο, με τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δικαιολογούν τη νέα ΚΑΠ. Και τέλος, θα αναλύσω τα διάφορα προτινόμενα μέτρα και τις ε, προτάσεις και συστάσεις ε, καθώς και τροποποίηση των μέτρων. Υπάρχει δηλαδή και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να γίνει από ακαδημαϊκής πλευράς. Το πρώτο θέμα Είχαμε πολλές ε, εκθέσεις και μας είπαν ότι η γεωργία ενέχει πολλούς κινδύνους. Δεν υπάρχει όμως κάποιος ε, ιδιάζων κίνδυνος που αφορά τη γεωργία. Κανένας κίνδυνος δεν αφορά αποκλειστικά τη γεωργία και πολλές φορές αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης και που οδηγούν στην αστάθεια. Δηλαδή η προσφορά και η ζήτηση ε, βραχυπρόθεσμα δεν επηρεάζουν τις ε, τιμές όταν υπάρχουν δραστικές αλλαγές από πλευράς προσφοράς ή ζήτησης τότε οδηγούμεθα στην αστάθεια. Πρόκειται για τον νόμο του Κίνγκ. Και αυτή η αστάθεια είναι ολέθρια από οικονομικής πλευράς δεν επιτρέπει από τους οικονομικούς φορείς να λάβουν τις σωστές αποφάσεις οικονομικής εμβέλειας. Γι' αυτό πολλές φορές μας λένε ότι η αγορά δεν θα φτάσει στη βέλτιστη δυνατή λύση, χρειάζεται η δημόσια παρέμβαση. Αλλά το θέμα είναι πιο δυσχερές, διότι υπάρχει πληθώρα μηχανισμών και γι' αυτό ο νόμος του Κίνγκ είναι ατελής. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί που ήδη υπάρχουν. Καταρχήν η αποθήκευση. Η αποθήκευση επιτρέπει την εξομάλυνση των τιμών. Δηλαδή αποθηκεύουμε όταν είναι χαμηλές οι τιμές και ε, βγάζουμε από τις αποθήκες όταν οι τιμές είναι υψηλές. Έτσι εξομαλύνονται οι διαφοροποίησεις των τιμών. Υπάρχει λοιπόν μια ασυμμετρία στην εξέλιξη των τιμών. Οι τιμές μπορεί να είναι χαμηλές, αλλά ποτέ δεν είναι απόλυτα, απόλυτα χαμηλές. Όλα σχετίζονται με την αποθήκευση. Επίσης το εμπόριο επιτρέπει να κατανείμουμε τους, ε, τους παράγοντες τυχεότητας Δηλαδή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε γεγονότα που ανακύπτουν στο νότο της Ευρώπης και όχι στο βορρά και τούμπαλιν. Δηλαδή, εάν η απόδοση των τιμών σιτηρών δεν είναι τόσο υψηλή, σε άλλες είναι, όπως στην Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ αλλά βλέπετε ότι διεθνώς η απόδοση των τιμών σιτηρών είναι ε, πολύ καλύτερη από τα μεμονωμένα στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν άλλες επιπτώσεις σε σχέση με τις μεμονωμένες χώρες και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές. Πέρα από τους ε, ε, μηχανισμούς της αγοράς που απαλύνουν τις ε, τιμές, που εξομαλύνουν τις τιμές, υπάρχουν και άλλοι οικονομικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για τις συμβάσεις και πολλές φορές λέμε ότι υπάρχουν συμβάσεις άναντι ή κάταντι, δηλαδή με τον αγροτικό τομέα ή τομέα τροφίμων ή με τις ασφάλειες με τους χρηματοοικονομικούς, τους θεσμικούς δηλαδή επενδυτές και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν συμβάσεις επιμερισμού των κινδύνων. Και δεν λέω ότι θα πρέπει να φτάσουμε στην επίμορτο αγροληψία όπως ίσχυε ε, σε παρελθόντες αιώνες, αλλά αυτό το σύστημα υπάρχει εν μέρη για να επιμερίσουμε τους κινδύνους μεταξύ του παραγωγού, του αγρότη, του παραγωγού της πρώτης ύλης και του, του, της άμεσης πηγής παραγωγής, δηλαδή της γης. Υπάρχει λοιπόν διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Δεν μιλάμε για μία δραστηριότητα, μπορούμε να έχουμε πληθώρα ε, δραστηριοτήτων. Δεν, μπορεί να παρά... δεν καλλιεργεί κανείς μόνο τομάτες, αλλά πολλά ο ποροκυπευτικών όταν ε, υπάρχει δυνατότητα. Επίσης, για να μειώσουμε τους κινδύνους θα πρέπει να ληφθούν επενδυτικές αποφάσεις όταν ε, δεν έχουμε καλές χρονιές, ε, μειώνονται οι επενδύσεις και το αντίθετο. Και επίσης οι αποφάσεις εξαρτώνται από τις αποταμιεύσεις και την πιστοληπτική ικανότητα. Δηλαδή τις κακές χρονιές στην κακή συγκομιδή χρησιμοποιούμε τις αποταμιεύσεις. Αυτό είναι ο νόμος του King. Δεν λέμε βεβαίως ότι οι μηχανισμοί αυτοί είναι τέλειοι. Κανένας δεν είναι απόλυτα θετικός. Δηλαδή υπάρχει το κόστος της αποθήκευσης. Τίποτα δεν χορηγείται δωρεάν. Υπάρχει το κόστος του εμπορίου, η μεταφορά των εμπορευμάτων. Τίποτα δεν χορηγείται δωρεάν. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσο οι δημόσιες αρχές μπορούν να μειώσουν ε, το κόστος των ε, μηχανισμών διαχείρισης των κινδύνων. Και υπάρχουν και οι ατέλειες της αγοράς. Υπάρχουν ε, τριών ειδών. Καταρχήν αυτές που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών. Μιλάμε για ασυμμετρίες ε, πληροφόρησης μεταξύ ενός ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου. Ε, ένας ε, ε, ασφαλιζόμενος πολλές φορές γνωρίζει ότι ο ασφαλιστής δεν ελέγχει το πλαίσιο. Γι' αυτό θα θέσει υψηλότερο ασφάλιστρο από αν γνώριζε τη συμπεριφορά του ασφαλιζόμενου και του τομέα του. Γι' αυτό το κράτος μπορεί να βοηθήσει για να διορθώσει αυτή την ασυμμετρία της αγοράς. Επίσης, ως προς το κόστος, η εσωτερική αγορά μπορεί να διαχειριστεί ε, τις τιμές, αλλά όχι όλων προϊόντων, διότι τα προϊόντα δεν είναι ομοιογενή. Άρα για το βόλιο κρέας δεν μπορούμε να ορίσουμε μια απόλυτα σωστή εσωτερική αγορά. Μας ε, ενδιαφέρει και επαλήθευση του προϊόντος. Και υπάρχουν και οι ε, ανασφάλειες, δηλαδή ότι ως προς τον νέο του Σμάλεμπεργκ κανένας δεν τον γνώριζε στο παρελθόν και δεν ήξερε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του. Εάν λοιπόν αυτά τα ε, γεγονότα, αυτά τα τυχαία γεγονότα ε, οδηγούν σε ατέλειες, αυτό το βλέπουμε στην ε, πράξη. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει δημόσια παρέμβαση άναντι η οποία υφίσταται τις διαφοροποιήσεις των τιμών. Μάλλον κάταντι και όχι άναντι. Άρα όλο το δίκτυο επιμερίζεται και επομίζεται τους κινδύνους, θετικούς ή αρνητικούς. Ένα δημόσιο αγαθό έχει σχέση με το ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή κάποιος θέλει να εμβολιάσει το ζωικό του κεφάλαιο. Θα πρέπει να δει τι επιρροές, τι εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν τον εμβολιασμό. Επίσης, η διαχείριση των καταστροφών είναι ένα άλλο θέμα που αφορά και έχει επιπτώσει και στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό προσπαθούμε να αναχαιτήσουμε τα αρνητικά στοιχεία των αγορών. Τι μας λέει τώρα η Κομισιόν, γιατί θα πρέπει η ΚΑΠ να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Γιατί όπως ισχύει και στην επίμορτο αγροληψία δεν ισχύει σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπως και η ασφαλιστική διαδικασία δεν είναι ίδια παντού. Γιατί στην Ευρώπη λοιπόν χρειαζόμαστε μία πολιτική διαχείρισης αγροτικών κινδύνων. Εδώ βασίστηκα στις μελέτες, στη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που συνοδεύει τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Η Επιτροπή αξιολόγησε τις τρεις εναλλακτικές που υποβλήθηκαν το 2010 και με βάση αυτή τη μελέτη αντικτύπων προσπαθούν προσπαθούμε, προσπαθεί η Επιτροπή να ορίζει πολιτικές αντιμετώπισης κινδύνων. Πέρα από τα επιχειρήματα που αφορούν το κάθε μέτρο χωριστά, υπάρχουν ε, δύο επιχειρήματα, ότι η αστάθεια των γεωρικών τιμών θα ε, αυξηθεί και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Κομισιόν, διότι αυτή η ιδέα είναι διαδεδομένη. Δεν ξέρω από πού προέκυψε. Όλοι λένε ότι οι τιμές αυξήθηκαν πρόσφατα, άρα θα αυξάνονται στο διηνικές. Πού ξέρουμε όμως ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιμές. Η Επιτροπή προβάλλει τρία επιχειρήματα για την αστάθεια των γεωρικών τιμών. Οι κλιματικές αλλαγές, ο συσχετισμός με τις τιμές ενέργειας, τα βιοκαύσιμα και το γεγονός ότι χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότεροι γεωργικές αγορές οι οποίες χρηματοδοτούνται βραχυπρόθεσμα. Ως προς τις κλιματικές αλλαγές κανένας δεν τις αμφισβητεί. Εάν υπάρχουν τυχαίοι παράγοντες θα υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια. Βεβαίως δεν έχουν διενεργηθεί πολλές μελέτες ε, για τον ορίζοντα 2015 2015-2020. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτός ο παράγωνας στάθειας, αλλά δεν ξέρουμε ότι η εμβέλεια θα είναι τόσο μεγάλη και κατά τα μελλοντικά έτη 15-20. Δεν έχουμε ε, πολλά ε, μέσα ελέγχου ως προς τον αλληλοσυσχετισμό των τιμών ενέργειας τιμών πετρελαίου με βιοκαύσιμα, αυτό εξαρτάται γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο τα ε, βιοκαύσιμα παράγονται υπό έλεγχο και κατά πόσο αιτιολογείται η αυξημένη τιμή του πετρελαίου. Όταν μιλάμε για ευελιξία, το ε, ζήτημα δεν είναι σαφές. Ίσως στο μέλλον οι βιομηχανίες παράγουν πολύ περισσότερο αλλά εάν μειωθεί η τιμή του πετραλαίου, ίσως παράγουν και λιγότερο. Άρα το να πούμε ότι οι τιμές ε, της ενέργειας θα οδηγήσουν στην αύξηση των αγροτικών τιμών, αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο. Ε, άλλοι σκέφτονται το αντίθετο. Τέλος, ως προς τον χρηματοοικονομικό τομέα, ε, λυπάμαι, αλλά είναι ένας τομέας ο οποίος δεν μας δίνει εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία για να ξέρουμε ότι θα, ότι θα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος ως προς την, ε, τις ημερήσιες τιμές ή τις, τους βραχυπρόθεσμους δείκτες ισχύει η αστάθεια των τιμών. Αλλά τώρα το να πούμε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να ε, αποφασίσουν ως προς την παραγωγή, του, δεν, παραγωγή τους δεν έχουμε στοιχεία. Έχουμε βραχυπρόθεσμες ε, αναλύσεις και άρα η απόφαση περί παραγωγής γίνεται μία φορά το χρόνο, δηλαδή η παραγωγή σύτου. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αλληλοσυσχετισμό των ημερησίων αναλύσεων και του ετήσιου ρυθμού παραγωγής. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να βάλουμε δεν μπορούμε να προβάλλουμε αυτό το επιχείρημα γιατί εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις βραχυπρόθεσμες αγορές για να διαχειριστούμε την αγορά. Αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα χρήση αυτών των μέσων με βάση τους ε, βραχυπρόθεσμους ε, δείκτες. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και αστάθεια, έμεση αστάθεια, δηλαδή καλύπτει κανείς τις ανάγκες με βάση τις εναλλακτικές που διαθέτει η, τιμή των εναλλακτικών μειώνεται, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αυξηθεί αναγκαστικά. Ένα άλλο επιχείρημα της Κομισιόν είπε ότι χρειαζόμαστε την ΚΑΠ γιατί τα εισοδήματα, τα αγροτικά εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά και ασταθή. Γιατί πέρα από τις γεωργικές τιμές υπάρχει και η αύξηση των, εσόδων και η συρρήκνωση της αγοράς. Εδώ και 15 χρόνια ακούμε αυτά τα επιχειρήματα. Δηλαδή κάθε φορά που μεταρρυθμίζουμε την ΚΑΠ γίνεται λογός για χαμηλά εισοδήματα και για συρρήγνωση αγοράς από το 1992 και μετά τα ίδια ακούμε. Ίσως, αλλά εδώ και 15 χρόνια δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άλλοι εμπειρογνώμονες που το αναφέρουν. Έχουμε στατιστικά στοιχεία εσόδων που απορρέουν από τη γεωργική δραστηριότητα, αλλά όχι έσοδα από τα γεωργικά νοικοκυριά. Γιατί κανείς μπορεί να ασχολείται και με άλλες παράπλευρες δραστηριότητες. Στην ιστοσελίδα της Κομισιόν ε, μας ε, αναφέρεται ότι εδώ και 15 χρόνια τα εισοδήματα από τη γεωργία μειώνονται δραστικά. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ και 15 χρόνια η τιμή της γης αυξάνεται συνεχώς. Πώς ε, μπορούμε να τα συμφιλιώσουμε όλα αυτά, δηλαδή χάνονται χρήματα αλλά επενδύονται και περισσότερα χρήματα. Ξέρω ότι το θέμα της εγγύου ιδιοκτησίας είναι περίπλοκο και αυτό ισχύει και για τη, και για τη Γαλλία όμως. Ε, υπάρχει ένα πλαίσιο διαχείρισης της εγγύου ιδιοκτησίας και έχει σημασία ε, που υπάρχει έγκυος ιδιοκτησία και που υπάρχει ε, ενοικίαση της γης. Ίσως πρόκειται για μία φούσκα της εγγύου ιδιοκτησίας, αλλά αυτές τις ε, φούσκες τις γνωρίζουμε εδώ και 15 χρόνια. Μιλάμε για αδυναμία, ίσως είναι υπαρκτή, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες απόδειξης. Και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Ένα άλλο επιχείρημα αφορά τη ε, μεταφορά των τιμών στην διατροφική αλυσίδα. Από μηχανιστικής πλευράς, εάν η τιμή κατανάλωσης είναι σχετικά σταθερή σε σχέση με την αγροτική τιμή, αυτό σημαίνει ότι η κεφαλαιακή απόδοση είναι σταθερή. Άρα ε, υπάρχει ε, μία αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των δύο. Έχει όμως σημασία να δούμε κατά πόσο στη μεταποίηση οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Δεν έχουμε πληροφορίες απόδειξης. Δείτε την έκθεση για το γάλα της ε, ε, ε, Επιτροπής υψηλόβαθμων εμπειρογνωμόνων για να δείτε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με την ε, βιομηχανία μεταποίηση και διανομή. Είναι δύσκολα μετρήσιμες αξίε, γιατί δεν πρόκειται για ένα προϊόν και ένα χρόνο. Πρόκειται για στοιχεία που πήρα από την Κομισιόν. Έχετε στο κόκκινο την τιμή που καταβάλουμε εάν είχαμε ε, βούτυρο σε σκόνη. Και βλέπετε στο μπλε την τιμή που καταβλήθηκε πραγματικά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση δηλαδή που θα μπορούσε να, να καταβάλει ο τομέας της βιομηχανίας, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Και βλέπετε ότι το 2008-2009 είναι το αντίθετο, ισχύει το αντίθετο. Αν δείτε από το 1 μέχρι το 7 έχασαν εκείνοι που παρήγαν βούτυρο σε σκόνη. Αν δείτε τα στοιχεία του 7, βλέπετε ότι υπάρχει ατέλεια στις τιμές, αλλά θα πρέπει να δούμε μακροχρόνια κατά πόσο γίνονται επενδύσεις οι οποίες ε, αποβλέπουν σε κάτι το συγκεκριμένο και αποδίδουν σε τα τελευταία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε τι κάνει, τι επιτυγχάνει ο άναντι τομέας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλώς χρειαζόμαστε πληροφορίες για τις επιμέρους διορθώσεις. Αυτά ως προς τα ε, επιχειρήματα. Τώρα, ας ε, δούμε τις προτάσεις και να δούμε πώς μπορούμε να τις ε, ε, διορθώσουμε. Υπάρχουν, υπάρχουν ε, πολλοί κανονισμοί για τις άμεσες επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις κινδύνου. Δηλαδή μιλάμε για διαχείριση κινδύνου. Έλαβα υπόψη όλους αυτούς τους επιμέρους, τους μίζονες παράγοντες και θα τους δω έναν έναν. Θα δω κατά πόσο είναι θεμητοί αυτοί οι παράγοντες σε σχέση με τα θεωρητικά οικονομικά. Η παρέμβαση που ισχύει στην ιδιωτική αποθήκευση δεν μιλάμε για μίζονες αλλαγές. Δεν λέω ότι δεν έχουν επέλθει καθόλου ε, αλλαγές στο σόργο και σε άλλα προϊόντα. Μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν έχουν επέλθει μίζονες αλλαγές στην ε, τιμή αναφοράς και τιμή παρέμβασης. Και ως προς την παρέμβαση, η παρέμβαση είναι υποχρεωτική για τρία προϊόντα. Για το σίτο, για ε, για το βούτυρο για το βούτυρο σε σκόνη και για το αποβουτυρωμένο γάλα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αποθηκεύσουμε και πότε θα βγουν αυτά τα προϊόντα από την αποθεματοποίηση. Η Κομισιόν πολλές φορές μας λέει ότι τη, ε, διαχειρίστηκε την κρίση του γάλακτος του 2009. Όταν δούμε όμως τις αντιδράσεις των άμεσα ενδιαφερομένων κατά τη διαχείριση της κρίσης του γάλακτος, δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη. Και αυτό το βλέπετε στην στήλη που αφορά το γάλα. Ως θεωρητική λοιπόν εμείς ε, έχουμε πληθώρα αμφιβολιών. Με συγχωρείτε, δεν φαίνονται οι διαφάνειες. Je... Donc, euh... Et euh, Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι η παρέμβαση σήμερα, όπως ορίζεται, αφορά περισσότερο ένα μέσο υποστήριξης των τιμών και όχι διαχείρισης κινδύνων. Και γιατί το λέω αυτό γιατί η παρέμβαση ορίζεται μόνο ως προς τα σιτηρά αυτόματα. Είναι ε, περίεργο. Έχετε εδώ μία γραφική παράσταση όπου βλέπετε ότι υπάρχει μία ε, προθεσμιακή αγορά για τα σιτηρά που είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Άρα ε, έρχονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και βλέπουν ότι διατρέχουν κινδύνους όπως προς τη τιμή της αγοράς οι τιμές της αγοράς είναι πλέον δραστήριες. Πρόκειται για το μόνο αγροτικό προϊόν όπου παραμένει η παρέμβαση. Αυτή η εσωτερική αγορά καλύπτει τους κινδύνους, δηλαδή ε, αν υπάρχει διαφοροποίηση 150 ευρώ ανατόνο και 200, τότε δεν έχει νόημα η τιμή παρέμβασης γιατί είναι 100 ευρώ τον τόνο. Άρα έρχονται στο συνεταιρισμό οι αγρότες και το διαχειρίζονται μόνοι τους στην εσωτερική αγορά. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η παρέμβαση είναι ένα μέσο διαχείρισης κινδύνων. Είναι ένα ιστορικό μέσον υποστήριξης των τιμών. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί η παρέμβαση δεν θα έπρεπε να αφορά όλα τα γεωργικά προϊόντα. Γιατί να μην ισχύει για τα ελαιούχα προϊόντα, γιατί ισχύει μόνο για τα σιτηρά, γιατί πρέπει να παίρνουμε ε, μόνο τα σιτηρά, γιατί υπάρχουν προϊόντα υποκατάστασης, γιατί να μην ισχύει στα ζαχαρότευτλα, στους ελαιούχους σπόρους και ούτω καθεξής. Και πολλοί θεωρητικοί ζητούν την απαλυφή εγώ όμως προτείνω να κρατήσουμε ένα μίνιμουμ παρέμβασης μακροχρόνια. Ακόμα και για τα σιτηρά, διότι κάποιος που θέλει να επενδύσει στην γεωργία το κάνει μακροπρόθεσμα. Άρα οι προθεσμιακές αγορές αφορούν μία, δύο ή τρεις συγκομιδές το πολύ, ενώ εδώ μιλάμε για 5, 10, 15 χρόνια. Δεν μπορώ λοιπόν να καλύψω την επένδυσή μου μέσα σε μία 15 ετία. Και η αγορά είναι πλήρης μόνο μακροχρόνια. Ενώ λοιπόν θέλουμε μακροχρόνια κάλυψη, τι μπορούμε να κάνουμε για τους αγρότες. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε κατά πόσο δούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρέμβαση. Υπάρχουν και θεωρητικές παρεμβάσεις, αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό που, από αυτό που έχουμε σήμερα. Έχω υποβάλει προτάσεις που θα συζητηθούν από τους συναδέλφους και πιστεύω ότι η τιμή παρέμβασης δεν μπορεί να είναι σταθερή. Αντίθετα, θα πρέπει να αναθεωρούνται οι τιμές παρέμβασης. Όμως χρειάζονται, χρειάζεται διαφάνεια ως προς κανόνες και το κόστος παραγωγής σχετίζεται με τις τιμές που προσμένουμε και τις σε την επένδυση σε γεωργικά προϊόντα. Δηλαδή προβλέπουμε τις τιμές Εάν ορίζουμε την τιμή παρέμβασης με βάση το κόστος παραγωγής, τότε θα φτάσουμε σε μια κάπ της δεκαετίας του 60. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ευέλικτες τιμές ανάλογα με την εξέλιξη των, της παγκόσμιας αγοράς και τιμών. Χρειάζεται λοιπόν εναρμόνιση μεταξύ τομέων και, και διαφάνειας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε μακροχρόνια. Ως προς τις ε, τομεακές επιδοτήσεις, μιλάμε για τα οποροκυπευτικά και τον αμπελοεινικό τομέα. Δηλαδή είχαμε τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του 2008 με λιγότερες άμεσες παρεμβάσεις, απόσυρση και διαχείριση των κινδύνων με βάση τα διάφορα ασφαλιστικά σχήματα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε αυτά τα μέσα για μία περίοδο καθαρά μεταβατική. Όπως είπα και για τις επενδύσεις, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες από σήμερα σε αύριο. Χρειάζεται μία μεταβατική φάση. Πόσο θα διαρκέσει εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα των επενδύσεων σε αυτό το τομέα αλλά αν αναθεωρήσουμε το 2008, το 2012 δεν έχουν αποσβεστεί οι επενδύσεις γενικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισχύουν στο δίνεκές Μακροχρόνια δεν έχουν ε, νόημα, διότι στο, στα προκυπευτικά πολλοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα. Και άρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τον ορίζοντα του 2020. Τώρα, ως προς τις συμβάσεις, το θέμα αυτό συζητήθηκε με το πακέτο του γάλακτος. Θα πρέπει να διευρύνουμε το επάγγελμα, τα επαγγέλματα αυτά. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ακόμα και οικονομικά τα διάφορα επαγγέλματα τη στιγμή που μιλάμε για σωστή οικονομική πληροφόρηση. Η οικονομική πληροφόρηση δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να καταβάλλεται ένα αντίτιμο. Όταν δεν υπάρχει εσωτερική αγορά, πώς μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στην αγορά. Άρα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αρκετούς τομείς. Άρα χρειάζεται δημόσια επιδότηση για την διάχυση και διάδοση πληροφοριών. Τώρα, να πούμε όμως τώρα ότι θα πρέπει να έχουμε διαπραγματευτική δύναμη σε όλη την αλυσίδα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί σε αυτή τη μετάβαση θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπτώσεις στην παραγωγή στη μεταβατική αυτή περίοδο. Και είχαμε πολλές αποφάσεις ε, των, ε, των αρχών ανταγωνισμού όπως στη Γαλλία. Η αρμόδια αρχή του ανταγωνισμού πάντα θα επεμβαίνει. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές και τον όγκο συναλλαγών. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετέχουν και να υφίστανται τις απόρριες του κινδύνου. Και βεβαίως μέσα στα πλαίσια των συνεταιρισμών αυτό γίνεται καλύτερο. Ως προς τις ανάγκες της αγοράς, νομίζω ότι έχω μείνει λιγάκι πίσω. Τι προτείνεται. Προτείνεται να κρατήσουμε τα μέτρα συναλλαγών. Βεβαίως ξέρω ότι γίνονται και στον ΠΟΕ αλλού διαπραγματεύσει επί του θέματος οι αποφάσεις των άλλων κρατών ε, δεν είναι σίγουρες. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει επέμβαση, αλλά δεν ξέρουμε πότε η Αργεντινή θα κλείσει τα σύνορά της ή πότε η Ρωσία θα κλείσει τα σύνορά της. Πρόκειται για μια πολιτική καθαρά απόφαση. Δεν χρειάζεται λοιπόν ένα ασφάλιστρο γι' αυτό. Όμως μπορεί να έχει επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές τιμές. Άρα θα πρέπει να αποφευχθεί. Άρα μέσα στα πλαίσια του αγροτικού λόμπι, των αγροτικών λόμπι, δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε εγχώριες αποφάσεις που διαλύουν την παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει να έχουμε αποτρεπτικά μέτρα έτσι ώστε άλλες χώρες να μην λάβουν μέτρα που ε, κυρώνουν, που ζημιώνουν όλες τις χώρες. Μπορεί να γίνει αυτό με δασμούς, με τέλη, πώς. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές μιλούσαμε για προϋπολογισμό που σχετίζεται με τα δεδομένα ΠΟΕ. Αυτό όμως τώρα δεν ισχύει, γιατί κάναμε ό,τι μπορούσαμε από τη δική μας πλευρά. Εάν οι άλλοι ε, καταβάλουν προσπάθειες, τότε θα σταματήσουμε τις επιδοτήσεις εξαγωγών. Αυτό αναφέρεται, αλλά είναι επιζήμιο πολλές φορές. Όταν διευρύνουμε το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε στη γεωργία. Όπως έχει το κείμενο δεν μπορούμε να απαλείψουμε τις επιστροφές κατά τις εξαγωγές. Αλλά αυτό δεν είναι καλό ε, σήμα. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ισχύει έτσι αυτός ο αποτρεπτικός χαρακτήρας. Είμαι υπέρ των ε, παρεμβάσεων σε σχέση με την φύση αυτών των ε, μέτρων, δηλαδή για ένα αποθεματικό προς την κρίση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνουν άμεσες καταβολές. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για για 3,9 δις ευρώ για το 14-20. Δεν ξέρουμε την εμβέλεια της κρίσης, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε δημοσιονομικά. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι απόρριες και τη στιγμή που δεν ξέρουμε την ε, εμβέλεια της ζημίας, δεν μπορούμε να ξέρουμε και την εμβέλεια της αντιστάθμισης. Και μετά βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να υφίστανται κυρώσεις και ζημία η γεωργοί. Έγινε μια προσωμείωση για τον αυθόδη πυρετό και δεν ξέρουμε κατά πόσο ζημιώνονται μόνο οι αγρότες. Μάλλον δεν σημειώνονται, δεν μόνο οι αγρότες αλλά και τα σφαγεία και ο μεταποιητικός τομέας και ούτω καθεξής. Ως προς τις ποσοστώσεις παραγωγής έχουμε το θέμα του περιορισμού των ποσοστώσεων. Ε, μιλάμε για την απαλυφή των ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης. Γνωρίζετε βεβαίως ότι η θεωρητική δεν είναι υπέρ των ε, ποσοστώσεων ζάχαρης. Μιλάμε για δημόσια αποθεματοποίηση και δεν ξέρω από ποια χρονική στιγμή ορίζουμε τις ποσοστώσεις. Πώς αποφασίζουμε να αποθεματοποιήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις ποσοστώσεις. Πότε είναι αρκετά υψηλή η τιμή έτσι ώστε να μειωθούν οι ποσοστώσεις παραγωγής. Εδώ δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Άρα δίνουμε τις ε, πληροφορίες, λέμε για συμμετοχή στις παγκόσμιες αγορές, αλλά αυτό δεν είναι ένα μέσο διαχείρισης κινδύνων. Μπορεί να είναι ένα μέσο εδαφικής συνοχής ε, ως προς την εδαφική παραγωγή, αλλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο. Είναι νέες οι πληροφορίες ως προς τον τομέα της ζάχαρης. Οι εκπρόσωποι ζήτησαν να αναβληθεί αυτή η απόφαση. Από ό,τι κατάλαβα, από τις πρόσφατες επενδύσεις σε αυτό το τομέα, μετά από την εφαρμογή της κοινή οργάνωσης αγοράς της ζάχαρης 2006-2007 ισχύει αυτό το καθεστώς και δεν μπορούμε να πούμε ότι έπεσαν οι τιμές, διότι η τιμή της ζάχαρης μετά από το 2006-2007 δεν ε, αναλώθηκε. Δηλαδή τα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα αρνητικά. Άρα η απόδοση των επενδύσεων δεν ήταν κακή. Άρα το να αναβάλουμε αυτή την απόφαση δεν είναι κάτι το σκόπιμο. Εντάχει προς τις άμεσες πληρωμές Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα δημόσια αγαθά και η χορήγησή τους, γι' αυτό υπάρχουν και οι άμεσες πληρωμές και μπορούμε να έχουμε συνοδευτικές πληρωμές σε περίπτωση δυσχεριών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι βασικές πληρωμές ε, δεν είναι σταθερές. Λέμε αυτό είναι το κονδύλι και μετά σκάβουμε, σκάβουμε, σκάβουμε και στο τέλος μένει κάτι που αφορά τις ε, βασικές πληρωμές, οι οποίες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τα δημοσιονομικά. Δεν καταλαβαίνω εάν οι άμεσες πληρωμές έχουν κάποια χρησιμότητα, γιατί δεν ε, υπάρχει εγγύηση για αυτές. Εάν υπάρχει, αν είναι αναγκαίες, τότε πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε. Ως προς τις συνοδευόμενες πληρωμές, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. είναι το ίδιο ισχύει αν ε, χρειαζόταν να έχουμε τέτοιου είδους πληρωμές, σε τι τιμή θα τις είχαμε θα περάσουμε πάλι στην κοινή γεωργική πολιτική της δεκαετίας του 60 από ω ε, ζήτησης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι καλώ δεν προτάθηκε αυτό. Ω προς το, στα μέσα της, ε, του δεύτερου πυλώνα υπάρχει ένα τμήμα συγχρηματοδότηση, ε, επιδοτήσεις και κεφάλαια για τις ασθένειες με ε, χρηματοδότηση 30%. Από το 2001 υπάρχουν ε, συνεχείς εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λένε ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, δεν θέλουμε τέτοιου είδους ε, ε, εγγυητικές επιδοτήσεις. Πώς γίνεται όμως τελικά να υπάρχουν τέτοιου είδους επιδοτήσεις, γιατί, γιατί απλώς μεταφέραμε την ευθύνη στους γεωργούς και τους λέμε εσείς πρέπει να έχετε τα μία αλληλοβοήθεια στα δικά σας. Είχαμε προτείνει και στο παρελθόν να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει για παράδειγμα στον τομέα του γυρινού κρέατος Είχαν πει τότε οι παραγωγοί θέλουμε μια μεγάλη επιδότηση με ένα, αλλά διαφορετικά δεν θέλουμε καθόλου. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος λοιπόν να μεταφέρουμε την ευθύνη στους, ε, στους παραγωγούς. Να ολοκληρώσω, αν και είναι δύσκολο κανείς να εξαγάγει συμπεράσματα, υπάρχουν πάντοτε κανόνες οι οποίοι δεν είναι σαφείς. Πρέπει να στείλουμε πολύ σαφή μηνύματα στους οικονομικούς ε, ε μπορούν να υπάρχουν ε, μέσα διαχείρισης κρίσεων. Γενικότερο συμπέρασμα επίσης είναι το γεγονός ότι η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη έλλειψη πληροφοριών για να δούμε την ποιότητα των επιχειρήσεων, να την αξιολογήσουμε και για να μπορεί ο κόσμος να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση για την κοινή γνώμη για να γνωρίζουν αν υπάρχουν προβλήματα, ανεπάρκειες κλπ. Και τέλος, τρίτο συμπέρασμα, κατά πόσο πρέπει να είναι στον πρώτο ή στο δεύτερο πυλώνα. Καταλαβαίνω ότι με τα δημοσιονομικά προβλήματα είναι περίπλοκα τα πράγματα. Δεν ε, πρέπει να μας διαφεύγει ότι έχουν μεγάλα περιθώρια ακόμη για τη διαχείριση κινδύνων τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν οι δημοσιονομικές πολιτικές και ε, υπάρχουν βέβαια και ε, και η έγκυος, η έγκυος ιδιοκτησία. Πάντοτε η έγκυος ιδιοκτησία είναι ένα σημαντικό κομμάτι και ένα σημαντικό παράγοντα. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίασή σας. Ήταν πάρα, πάρα πολύ λεπτομερής πολύ λεπτομερής και η παρουσίαση των προβλημάτων ε, που έχουμε. Σας άφησα χρονομιλίας γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για μας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια ομάδα επισκεπτών που παρακολουθεί τις εργασίες μας σήμερα από την Πορτογαλία. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά. Είναι μια ομάδα ε, της Ένωσης ε, Γεωργών της Πορτογαλίας. Να αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Ο κύριος Άγνιου είναι ο πρώτος ε, ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι θα καταλάβετε, φαντάζεστε ότι δεν συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Εγώ είμαι γεωργός και αν δει κανεί το πρώτο νήμα τη παρουσίαση, είναι σαν να προσπαθείτε να πάρετε όλο τον κίνδυνο από του Γεωργιαίου και να τον μεταφέρετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό και είδαμε τι έγινε. Ε, για παράδειγμα, στη Σοβιετική Ένωση. Εγώ είμαι πρόθυμος να αναλάβω κίνδυνο και υπάρχουν χιλιάδες ε, τρόποι να μπορέσουμε να, το, ε, να τον αναλάβουμε αυτόν τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, οι πωλήσει Τα futures είναι πραγματικά ένας πολύ καλός τρόπος. Μπορεί κανείς ε, να το κάνει αυτό τώρα ε, με κάποιο τίμημα, δεν λέω, αλλά μπορεί κανείς να αγοράσει την επιλογή του να πουλήσει και αυτή είναι μια, του να πουλήσει. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ε, επιλογή για τους γεωργούς. Καλό είναι και οι συνεταιρισμοί, αλλά ο ιδιοκτήτη του συνετορισμού μπορεί να αποφασίσει τι θα πουλήσει ε, και τι δεν θα πουλήσει. Οπότε υπάρχει μία εξισορρόπηση. Είπατε στην παρουσίαση ότι οι συνεταιρισμοί, κατά τη γνώμη σα, είναι πάρα πολύ ισχυροί. Αυτό εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Γιατί όντω, ε, αν ήταν ισχυρότεροι, αυτό θα βοηθούσε του γεωργού. Υπάρχει και ένα ακόμη τρόπο, ειδικότερα στον τομέα της ε, Εντατική κτηνοτροφίας ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, ε, κάποιο είδου διαφορετική χρηματοδότηση γιατί μπορούν να αναλάβουν έναν κίνδυνο κάπως περισσότερο μοιρασμένο. Και δεν νομίζω ότι μπορεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει περισσότερο σε αυτό. Ρωτήσατε επίση για το θέμα των τιμών ε, της γης. Δεν μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο πέφτουν οι τιμές και για ποιο λόγο ενώ πέφτουν οι τιμές εγγύου ιδιοκτησία αυξάνονται οι τιμές, ε, ότι υπάρχουν διάφορε, διάφορα είδη φορολόγηση, ε, υπάρχει επίσης η ανακούφιση με rollover, με μεταφορά κονδυλίων, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά μα είπατε. Αν οι γεωργοί δεν βγάζουν το ψωμί τους με αυτές τις Υψηλέ τιμέ των αγαθών, για ποιο λόγο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν όλα, να τα θέλουν όλα. Υπάρχει Επίσης, ε, όσον αφορά τις τιμέ παρέμβαση, από ό,τι κατάλαβα, ο η διαφωνεί απολύτω με αυτά που είπατε και γι' αυτό χρειάστηκε να σταματήσουμε να το κάνουμε και διορθώστε με αν κάνω λάθο. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις ζάχαρης που τελειώνουν το 2015, κατά τη γνώμη μου για το Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον πάνε πολύ γρήγορα τα πράγματα έπρεπε να κλείσουμε πριν από 3-4 χρόνια τις ε, εγκαταστάσεις παραγωγής σε ζάχαρης ε, και το να τις ξανανοίξουμε δεν είναι δυνατόν σε δύο χρόνια. Ε, οπότε σας ζητούμε μία καθυστέρηση, διαφορετικά το Ηνωμένο Βασίλειο θα πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, για τους, στους, στον, στον τομέα αυτών της, και, τον, και τον τομέα του ζαχαροκάλαμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέσατε πολύ σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τον τομέα της ε, ζάχαρης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιαζεμπού. Ε, και μετά... Ε, Alors, euh, je Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Χωσέ Βέ, Συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό σε άλλες γλώσσες στη Γαλλία θα ήμουν ε, σήμερα ε, μεταξύ των ε, γεωργών που είναι θαμένοι λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων. Μας αναφέρατε τα πάντα, ακόμα και για την οικονομία της γεωργίας μιλήσατε και μιλήσατε και για τη λογική της οικονομίας που πρέπει να αναπτυχθεί στη γεωργία. Ένα ερώτημα λοιπόν μου γεννιέται, όχι τόσο στον ε, ομιλητή μας, γιατί έχει, να, έχει το δικαίωμα να πει ό,τι ε, πιστεύει και ε, δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για την, στην οποία πρέπει να συζητήσουμε για τα εργαλεία της κοινή γεωργικής πολιτικής διαφορετικά. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε ένα εργαστήριο ε, πλουραλιστικό που θα ακούγονταν όλες οι απόψεις, αλλά εδώ μιλάμε για, ε, τελικά για, μια, για, για το ένα εργαλείο πίσω από το άλλο ε, καταλαβαίνω ότι μπορούμε να έχουμε ένα γεωργικό μοντέλο χωρίς αγρότες, χωρίς γεωργούς, που δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα κοινωνικά ζητήματα, τα πολιτισμικά ζητήματα, ε, την ιστορική σχέση ε, που έχει η γεωργία με τα, τις χώρες μας. Ε, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ένα, ε, ένα, μια θεώρηση των πραγμάτων με πολύ αφηρημένες έννοιες όπου δεν θα συμμετέχουν καθόλου οι γεωργοί. Δεν ξέρω ούτε έναν γείτονα που δουλεύει στον υπολογιστή για να μπορέσει να πουλήσει ή για να μπορέσει να ε, κυκλοφορήσει, να διαθέσει τα προϊόντα του στην αγορά για να μπορέσει επίσης να χρησιμοποιήσει συστήματα προστασίας μέσω του υπολογιστή. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν μιλάμε για έναν μεγάλο μάνατζερ, ενδεχομένω να μπορεί να γίνει, αλλά στην πραγματικότητα τι ποσοστό της γεωργίας είναι σήμερα στην Ευρώπη αυτό. Λέμε σήμερα πώς είναι δυνατόν να διατηρήσουμε μια γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πραγματικούς γεωργούς και πώς είναι δυνατόν να διατηρήσουμε την, ε, ε, τη γεωργία και τους γεωργούς. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε το δικό σας μοντέλο. Μας λέτε σήμερα για παράδειγμα ότι είστε υπέρ του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Προφανώς έτσι ανοίγουμε τις αγορές και αν υπάρχει ένα πρόβλημα με το Μερκοσούρ, με τον Καναδά ή την Ινδία, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θα μα βοηθήσει, όπω βοήθησε και του εργαζομένου στο Βιλβόρμπι ή τη ε, Μιτάλ που του απολύσαμε γιατί ε, πρέπει να κλείσουν ε, οι επιχειρήσει γιατί δεν έχουν πια κέρδο. Αυτό λοιπόν το ερώτημα που μου δημιουργείται σήμερα είναι το εξή δεν ε, υπάρχει μία ευρεία θεώρηση της γεωργίας, έχουμε μία οικονομική στική για να το πω έτσι, με λίγο βάρβαρους γλωσσικούς όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ε, βλέπω να λύνουμε το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και δεν θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτό το όραμα, το οποίο είναι πολύ ε, τμηματικό, πολύ κατακαιρματισμένο, γιατί ξέρετε, είστε οικονομολόγος, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα ακούσουμε χιλιάδες λόγους, χιλιάδες ομιλίες, είτε για, το, για την αντικυκλική ε, διαδικασία των πραγμάτων, είτε για τη διαχείριση της παραγωγής, ε, ε, είτε για το που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τις συνέπειες του οικονομικού μοντέλου της γεωργίας το ερώτημα μπορούμε, μπορεί να τοθεί και αλλιώ. Πώ είναι δυνατόν να προλάβουμε την κατάσταση ώστε να μην φτάσουμε στη διαχείριση κινδύνου. Δεν είμαστε υπέρ μια πολιτική που καλύπτει του κινδύνου, αλλά που του προλαβαίνει. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε για παράδειγμα για το γάλα τι έγινε με τις ποσοστώσεις γάλακτος παρά το γεγονός ότι δεν ήμουν μεγάλος θαυμαστής και υπερμαχός τους. Εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο συνολικής διαχείρισης όταν δούμε τη μακροχρόνια περίοδο των ποσοστώσεων αυτών υπάρχει εξίσωση σε σχέση με τους όγκους, υπήρχε μία σταθερότητα και μία κανονικότητα των τιμών. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ε, ε, λογική. Σήμερα το να λέμε απλώς, ε, απλώς διάλυση των πάντων είναι μια ιδεολογική επιλογή. Και εγώ βρίσκω απαράδεκτο σήμερα να δίνουμε το λόγο μόνο σε ένα συγκεκριμένο άτομο το, που μας λέει ότι είμαι εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινώσεων. Εγώ, διαφορε... εγώ διαφωνώ καθέτος με το συγκεκριμένο ε, για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πραγματικά βρίσκω αξιολύπητα αυτά που μας είπατε, αλλά σας σέβομαι γιατί έχετε το δικαίωμα να τα εκφράσετε. Ευχαριστώ πολύ. E, proszę o zabranie głosu panią poseł Brittę Reimers, następnie pan Michel Dante. Κύριος Ράιμερς έχει το λόγο. Η κυρία Ράιμερς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, εισηγησή σας και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που και εγώ τα βλέπω ε, με τον ε, ίδιο τρόπο. Έχω μία ερώτηση. Είπατε ότι ελάχιστες, ε, ελάχιστα δεδομένα είναι διαφανή και γνωστά. Τώρα, αν οι ε, γεωργοί αρχίσουν να διαπραγματεύονται για τις τιμές των προϊόντων, Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουν. Εκείνο όμως που γνωρίζουν πάντα είναι το σχετικό ύψος των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν. Εσείς λοιπόν τι πιστεύετε, είναι δυνατόν οι άμεσες ενισχύσεις να έχουν ε, αρνητική επίπτωση στις ε, τιμές αγοράς και πώλησης. Είναι δυνατόν οι ενισχύσεις ε, να έχουν και άμεσες επιπτώσεις στην έγκυο ιδιοκτησία. Είναι δυνατόν να υπάρχει τελικά και αρνητική επίπτωση στα εισοδήματα των γεωργών, διότι τα τελευταία 15-20 χρόνια που στηρίζουμε τη Γεωργία με τις άμεσες ενισχύσεις δεν κατορθώσαμε να σταθεροποιήσουμε ή να αυξήσουμε το εισόδημα των Γεωργών. Δεν κατορθώσαμε δηλαδή να επιτύχουμε τη σταθερότητα στην αγορά. Άρα δηλαδή προκλητικά, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, μπορεί κανείς να πιστεύει ότι οι άμεσες ενισχύσεις ε, είναι ε, λόγος ε, για το ότι επηρεάζονται οι γεωργοί στις διαπραγματεύσεις τους. Μερικές φορές τους λένε ότι θα λάβεις άνεσες ενισχύσεις αν πουλήσει ή αν διαπραγματευτείς την αγιοδιοκτησία. Κάνε μας κάποια καλύτερη τιμή, κάνε κάποια έκπτωση. Είναι δηλαδή δυνατόν ο γεωργός τις, ε, τις άμεσες ενισχύσεις του να τις καταβάλει σε διάφορους ε, και κατόπιν τούτου αυτό να επηρεάζει αρνητικά το εισόδημά του. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει άμεσα να γνωρίζω πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το θέμα. No ciekawe to, co Pani powiedziała, dlatego że dotychczas było tak, że w przypadku dopad bezpośrednich do produkcji Πολλές φορές οι άμεσες πληρωμές οδηγούν σε αλλαγή τιμών, δηλαδή συμπιέζονται προς τα κάτω οι τιμές ανάλογα με το γεωργικό είδος, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίστροφο. Άρα αυτό που θα έχει σημασία θα ήταν να βοηθήσουμε τους γεωργούς ως προς τα έσοδά τους. Στη συνεδρίασή μας ε, συμμετέχουν και βουλευτές από διάφορες χώρες, τους οποίους και καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας. Θα θέλαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι να μας πούν από ποια χώρα προέρχονται, από ποια οργάνωση όταν λαμβάνουν το λόγο, για να ξέρουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους δίνω το λόγο στον επόμενο βουλευτή. Merci. Bon, je voudrais... Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Ντόντε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ποιότητα κυρίω της παρουσίασή του τον ομιλητή, παρά το γεγονό ότι ο καθένας μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με αυτά που είπε. Είπατε κάπως εμέσως ε, αλλά ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε στις δημόσιες αρχές ε, την ε, δυνατότητα εξασφάλισης της αφήνειας της πληροφορίας, της πληροφόρησης. Δηλαδή πιστεύετε, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν έχει κανέναν άλλο ρόλο να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας, ε, εκτός από τη διαχείριση των τιμών και τη ρύθμιση των αγορών. Η... Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Πιστεύετε ότι η οργάνωση του κλάδου ε, από, την, ε, από το γεωργό μέχρι τους υπόλοιπους επαγγελματίδες του κλάδου Πιστεύετε ότι έχει κάποιο ρόλο εκεί ε, το δημόσιο τομέα και αν ναι, σε ποιο βαθμό και για ποιο λόγο. Dziękujemy pan poseł Hausnik, bardzo proszę i następnie pan poseł e, Κοιτάξτε, πιστεύω ότι εδώ έχουμε κάτι που ακούστηκε πολλές φορές ε, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, ε, δεν δίδονται συγκεκριμένε απαντήσεις και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί σε όλα αυτά τα θέματα να ακούμε ένα και μόνο εμπειρογνώμονα με μία ε, προκατηλημένη άποψη, γιατί δεν ακούμε περισσότερους. Ε, δεν πρέπει να ακούμε μόνο έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος δεν εκφράζει την άποψη της ε, πλειοψηφία. Αυτό που με εξέπληξε είναι αυτό που είπατε ότι πρέπει ακόμα να γίνουν πολλές έρευνες, να συγκεντρωθούν πολλές πληροφορίες. Ίσως για στο μέλλον να πρέπει να το κάνετε αυτό, αλλά όταν είπατε ότι δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ε, για κερδοσκοπίε στην αγορά, εκεί επιτρέψτε μου να βάλω εγώ ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τη στιγμή που ακόμα και ο Γάλλος ε, πρόεδρος είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεν είναι δυνατόν να λέει κανείς, δεν έχουμε αρκετές πληροφορίε Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ουσιαστική κερδοσκοπία στις ε, τιμές ε, των αγορών ε, βλέποντας ποια ήταν η κατάσταση και πώς εξελίχθηκαν οι τιμές. Δηλαδή η ζήτηση και η προσφορά δεν έχουν καμία σχέση με την εξέλιξη των τιμών. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην αγορά που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία αλλά είναι κερδοσκόποι και αυτούς πρέπει να τους απομονώσει η ε, πολιτική, όχι μόνο η γεωργική μεταρρύθμιση και κάτι άλλο. Είπατε ότι δεν ξέρουμε ε, κατά πόσο οι εξελίξεις ε, στις τιμές των καυσίμων ε, θα επηρεάσουν τη γεωργία. Και σε αυτό βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν δείτε λιγάκι την εξέλιξη της ε, τιμής των ε, τροφίμων, αν δει κανεί την τιμή του σιταριού, το σιτάρι, η τιμή του σιταριού ακολουθεί την τιμή του πετρελαίου περίπου με την ίδια ανωδική τάση. Είναι η ίδια καμπύλη. Άρα δηλαδή σαφώς υπάρχει σχέση ανάμεσα στην τιμή του πετρελαίου και στην τιμή του σιταριού. Και έχει και άμεση σχέση και με με την παραγωγή βιοκαυσίμων που λέτε ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα και αυτό με εξέπληξε. Επίσης είπατε ότι και η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει την κατάσταση. Ε, κοιτάξτε, πρέπει να δείτε τι κάνουν οι μεγάλες ε, ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, έχουμε μια μεγάλη αντασφαλιστική εταιρεία στο Μόναχο η οποία λέει ότι ειδικά στον γεωργικό τομέα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στην, στις αποζημιώσεις καταστροφών που έχουν άμεση σχέση με την κλιματική κλιματική αλλαγή. Κατόπιν είπατε ότι δεν επηρεάζουν οι κερδοσκόποι ε, της, ε, την αξία της γης. Βεβαίως ε, και στον γεωργικό τομέα εμπλέκονται πολλοί επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία, απλά επενδύουν στην γη ως αξία, ως αξία γης Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό οδηγεί σε εκτόξευση των τιμών γιατί όπως σας είπα εμπλέκονται άνθρωποι που είναι κερδοσκόποι. Επίσης αναφέρθηκε ότι ε, δεν είναι δυνατόν ε, να προβλέψει κανείς με σαφήνεια ε, το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στην Ευρώπη. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας. Νομίζω αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στην τιμή του γάλακτος. Αν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας στο γάλα στα 20 cent. Αυτό είναι περίπου κάτω από το ίμιση του κόστους παραγωγής ε, των παραγωγών. Δεν είναι δίχτυ ασφαλείας, είναι έσχατη βοήθεια, αλλά αυτό αυτό δεν έχει καμία σχέση. Επίσης, ε, στην ομιλία σας δεν ασχοληθήκατε τόσο με τη Γεωργία, αλλά νομίζω ότι με την ε, ομιλία σας είπατε περισσότερο ότι ναι, ε, πρέπει να απελευθερώσουμε τα πάντα και το σημαντικότερο είναι να είμαστε ανοιχτοί και να υπάρχει διαφάνεια στις αγορές, που δεν υπάρχει όμως και που πρέπει να την επιφέρουμε γιατί οι τιμές δεν προσανατολίζονται στο πραγματικό κόστος, όπως σας είπα υπάρχει τεράστια κερδοσκοπία. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, το ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και πρέπει να είναι στις ε, σκέψεις μας. Νομίζω ότι η γεωργία δεν είναι ένας ε, τομέας που μοιάζει με όλους τους άλλους ε, τομείς πρώτων υλών αλλά ειδικά στη Γεωργία χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο πλαίσιο. Ε, αυτό αποδείχτηκε ότι όταν υπήρξε ρύθμιση στις αγορές, είτε στο γάλα, είτε στη ζάχαρη, είτε στο κρασί, ε, προέκυψαν πολύ λιγότερες διακυμάνσεις και πολύ πιο ισόρροπες αγορές. Ε, πολύ μικρότερη αστάθεια από προϊόντα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε διεθνείς αγορές. Πολύ ωραία ο κύριος Φάιμον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Στην σημερινή εποχή σκεπτόμαστε πώς ακριβώς θα δημορφωθεί η κοινή γεωργική πολιτική στο μέλλον και ως εκπρόσωποι της Γεωργίας σκεπτόμεθα διάφορα πράγματα. Ετέθη το ερώτημα της ρύθμισης της αγοράς ζάχαρης. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώσαμε ότι εκτοξεύτηκε στα ύψη η τιμή της ζάχαρης. Οι καταναλωτές λένε ότι το πρόβλημα οξύνεται, ότι κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα ε, πολλοί επενδυτέ ε, είναι πρόθυμοι εκ νέου να επενδύσουν στη ζάχαρη με νέα δηληστήρια. Αλλά λόγω του συστήματος των ποσοστώσεων κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι το όλο σύστημα της ζάχαρης ε, πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Και τίθεται το ερώτημα, εσείς πώς το σκέπτεστε αυτό, συγκεκριμένα για τη ζάχαρη, τι έχετε να προτείνετε. Μπορείτε να σκεφτείτε μια μορφή ήπιας ε, χρηματοδότησης στο μέλλον, το τόσο σημαντικό αγαθό πώς πρέπει να προχωρήσουμε και πώς ε, μπορεί να γίνει η προσαρμογή στην, ε, στην παγκόσμια αγορά. Εγώ ε, συμφωνώ βέβαια ότι τα εργαλεία ε, βοήθειας που χρησιμοποιούμε πρέπει να περιοριστούν και ότι αυτά μπορούν να επηρεάσουν μόνο σε κάποιο βαθμό τη σταθερότητα της αγοράς γιατί οι άμεσες πληρωμές πράγματι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και μετά το 2013 οι πληρωμές αυτές θα είναι νομίζω οι ίδιες για το σύνολο των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερωτώμεθα όμως κατά πόσον ε, θα υπάρξει πιο δίκαιο ανταγωνισμός, κατά πόσον μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και θα υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Κύριος Άλβε, αυτή τη στιγμή αναλύουμε μία νέα κοινή οργάνωση της αγοράς και κινούμεθα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για αυτή την περίοδο που αρχίζει τώρα, το 2013. Μιλάμε για την αστάθεια των ε, τιμών, αλλά μιλάμε και για άλλες προκλήσεις, όπως η αστάθεια παραγωγής, η αύξηση του κόστους, που δεν ήταν ε, τόσο μεγάλη στο άμεσο παρελθόν, τη διατροφική ασφάλεια, την ανασφάλεια ως προς τις, τους μακροοικονομικούς παράγοντες, δηλαδή πιστοληπτική ικανότητα και ούτω καθεξής. Και η Επιτροπή προσπαθεί να ορίσει ένα δίκτυο ασφάλειας ή εξασφάλισης. Παράλληλα όμως μιλάμε για τον τομέα του γάλακτος και της ζάχαρης, όπου δεν ε, υπάρχει τόσο οργανωμένη αγορά και θα ήθελα να σταθώ στον τομέα του γάλακτος γιατί από ό,τι φαίνεται το 2013 θα ε, διαλυθεί αυτός ο τομέας. Δηλαδή μιλάμε για μια παραγωγή η οποία θα πολλαπλασιαστεί επί πέντε για χώρες όπως η Πορτογαλία. Και αν λάβουμε υπόψη την παρούσα ε, συγκυρία όπου έχουμε αύξηση κόστους, θα μειωθούν δραστικά οι τιμές. Άρα στα πλαίσια των, του υψηλότερου κόστους και χαμηλότερων ε, τιμών θα συρρυκνωθεί η, η αγορά. Δηλαδή υπάρχει περιορισμός περιθωρίων που θα έχει εδαφικές επιπτώσεις, διότι οι ποσοστώσεις ορίζονται εδαφικά. Και στην περίπτωση της Πορτογαλίας και άλλων χωρών δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε από αυτήν την συρρήκνωση, την μείωση των τιμών και ούτω καθεξής. Αυτή είναι και η ερώτησή μου. Αυτή η τομεακή προσέγγιση δεν θα πρέπει να είναι ίδια με την εδαφική, τη γενικότερη εδαφική. Σε σχέση με την χρηματοδότηση επίσης, μιλάμε για το γεγονός ότι δεν βασίζεται στην αστάθεια των τιμών. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα ισχύει η πρόσβαση στα μεγάλα ταμεία. Τι θα γίνει με την αγορά παραγόγων. Γιατί η, τη στιγμή που θα διαπραγματευόμαστε με χρηματοπιστωτικούς ογκόληθους, πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν θα υπάρχουν κλειδονισμοί στις τιμές για αυτούς ακριβώς που θέλουν να ορίσουν τις, τιμές, τις αγορές των παραγωγών, των παραγόγων συγγνώμη, για να μπορέσουν να ορίσουν τις τιμές. Πώς ε, να μην αποφύγουμε την κερδοσκοπία στην αγορά παραγόγων. Αυτό θα ήταν ολέθριο για την αγορά και για παρόμοια ταμεία τα οποία δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της αγοράς. Θα πρόκειται δηλαδή για μια συνεχιζόμενη ε, κερδοσκοπία. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Λουίς, Λουίς Κάπολας ε, Σάντος και μετά Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίαση του θέματος και σας ευχαριστώ για, ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ε, σύμφωνη γνώμη ή όχι. Όλοι ζούμε σε μια εποχή αστάθειας των αγορών, των τιμών και ανασφάλειας για τους γεωργούς με βάση την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Έχουμε να κάνουμε με μια απορριθμισμένη παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά διέπουν την αγορά. Και η αγορά ορίζεται και από παράγοντες που δεν ορίζονται, δεν ελέγχονται, όπως οι κλιματικές αλλαγές, όπου αντιμετωπίζουμε μεγάλη ξηρασία, όπως στη χώρα μου, και γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας ε, μηχανισμός υποστήριξης. Άρα το ζήτημα που τίθεται είναι ε, κατά πόσο μέσα στα πλαίσια μιας νέας ΚΑΠ θα θέλαμε να έχουμε ένα δίκτυ ασφαλείας που να επιτρέπει στους γεωργούς να προωθούν τη δραστηριότητά τους με ηρεμία. Κατά την άποψή μου, στις προτάσεις της Επιτροπής δεν υπάρχει αυτό το δίκτυ, γιατί έχουμε μία λίστα, έναν κατάλογο μηχανισμών και μέσων που δεν μας δίνουν τίποτα το καινούριο. Μιλάμε για τα μέσα που γνωρίσαμε και στο παρελθόν και υπάρχει και ένα σύνολο κανόνων το οποίο ε, σύνολο είναι άχρηστο. Θα γίνει και αυτή η συζήτηση. Μιλάμε για μία σειρά νέων μέσων που από πλευράς παρουσίωσης και συλλογιστικής δεν έχει νόημα. Όταν θέλουμε να δούμε έμπρακτα πώς ε, ε, ε, εφαρμόζονται, έχουμε πολλές αμφιβολίες. Θα ήλπιζα λοιπόν να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για τα νέα αυτά μέσα ή νέες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να εγγυηθούμε αυτό το δίκτυο ασφαλείας. Αλλά το θέμα αυτό είναι καθαρά πολιτικό και εμείς λαμβάνουμε τις πολιτικές αποφάσεις. Χωρίς πολιτικές αποφάσεις δεν θα μπορέσουμε να προβούμε στις ε, σωστές επιλογές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πολιτικό ε, δόγμα που ίσχυσε μετά από την ε, πτώση του τείχους του Βερολίνου. Μιλάμε δηλαδή για μια φιλελεύθερη προσέγγιση και απορρίθμιση και δεν μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή τη λογική στον ε, τομέα της γεωργίας. Θα πρέπει όμως να το κάνουμε και είμαι στη διάθεση του κυρίου Νταντά για να συζητήσουμε για τους δύο αυτούς πυλώνες έτσι ώστε να υπάρχουν μηχανισμοί που να παρεμβαίνουν στην αγορά και να μην μιλάμε για ένα κατάλογο ευσεβών πόθων που έχουν ε, αμεληταία αποτελέσματα. παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία πλειοψηφία στο Συμβούλιο, μία ε, φιλελεύθερη πλειοψηφία, εγώ βλέπω ότι οι ίδιοι ζητούν να παραμείνουν οι ποσοστώσεις για τη ζάχαρη. Δηλαδή είμαστε επιλεκτικά φιλελεύθεροι, φιλελεύθεροι για μερικά, αλλά παρεμβατικοί για άλλα. Δηλαδή είμαστε παρεμβατικοί για αυτό που μας αρμόζει τομεακά, όπως η ζάχαρη. Νομίζω λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, της γεωργίας και η επιτυχία μας βασίζεται σε μηχανισμούς που οδήγησαν σε ηρεμία και ασφάλεια. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτούς τους μηχανισμούς που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω ανασφάλεια για το μέλλον και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους μηχανισμούς και πώς μπορούν να αποτιμηθούν σωστά. Ευχαριστούμε Λουίς. Πατράου Νέβες. Και μετά ο κύριος ε, Γιάρ. Η κυρία Πατράου Νέβες. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εισήγηση, γιατί αποτελεί έναυσμα συζήτηση. Βεβαίω η αστάθεια των τιμών είναι ένα θέμα ύψη της σημασίας και είναι και αποφασιστική σημασία για το μέλλον. Εάν δεν καταπολεμήσουμε την αστάθεια των τιμών, δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις συγκεκριμένες παραγωγές και δεν θα μπορέσουμε να δελεάσουμε τους νέους έτσι ώστε να ε, ακολουθήσουν αυτό τον ε, επαγγελματικό προσανατολισμό. Όπως ήδη ελέγχθη, δεν υπάρχουν καινοτόμα στοιχεία από την Επιτροπή και το θέμα του, του δικτύου ασφαλείας, του δικτύου ασφαλείας δεν ε, αρκεί γιατί δεν υφίσταται. Έγινε λόγος για την ξηρασία στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και βλέπουμε ότι ακόμα και μεταξύ χωρών, εδώ μιλώ για την Ισπανία και την Πορτογαλία, για την Ιβυρική Χερσόνησο, δεν ξέρουμε πώς να ε, καταπολεμήσουμε την ε, ξηρασία τη στιγμή που δεν υπάρχουν και ασφαλιστικά προγράμματα όπως ισχύουν στην Ισπανία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κοινό κοινούς παρονομαστές, διότι βλέπουμε ότι η γεωργία ολοένα και απελευθερώνεται, είναι ολοένα και πιο ανταγωνιστική, αλλά δεν έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού. Και γι' αυτό ε, προωθείται αθέμητος ανταγωνισμός εξ αρχής. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όταν μιλάμε για τη γεωργία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν μιλάμε για οποιαδήποτε ε, δραστηριότητα. Μιλάμε για βασικά αγαθά που έχουν ε, μεγάλη σημασία. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την οικονομίστικη προσέγγιση. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η παραγωγή γεωργικών αγαθών αποτελεί ένα στρατηγικό μέσο Εάν έχουμε ε, αυτή την προσέγγιση, την οικονομίστικη προσέγγιση, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Γιατί υπάρχουν και άλλα μέρη του κόσμου που γνωρίζουν πολιτική αστάθεια και θα βρεθούμε στα χέρια άλλων, θα εξαρτώμεθα από άλλους. Εάν λάβουμε υπόψη τα διάφορα κράτη-μέλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γεωργία έχει μία πολυλειτουργικότητα, την οποία δεν ελέγχουμε πάντα. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να παρέμβουμε στα λογιστικά παραγωγής των δημοσίων αγαθών, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε γεωργία μόνο για ορισμένα κράτη-μέλη και όχι για άλλα, γιατί η γεωργία είναι υπεύθυνη όχι μόνο για την παραγωγή αγροτικών αγαθών, αλλά και για δημόσια αγαθά, για τον ε, ε, ορισμό, για τον προσδιορισμό των αγροτικών ε, πληθυσμών και ούτω καθαξής. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αμελήσουμε αυτή την αγορά. Κάθε φορά που μιλάμε για οικονομικά πρότυπα που ισχύουν για τη γεωργία θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς γιατί δεν μιλάμε για οποιοδήποτε τύπο οικονομικών αγαθών. Μιλάμε για είδη άμεσης ανάγκης, είδη επιβίωσης και γι' αυτό θα πρέπει να εξισορροπήσουμε εδαφικά τα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ρόλος μας εδώ είναι να εγγυηθούμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2013, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών και των περιφερειών. Και η, οικονομισ... οικονομιστική προσέγγιση βλέπει μόνο αριθμητικά στοιχεία απομονωμένα και βλάπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως προς τη συνοχή της και την ε, ανανέωσή της καθώς και την αντιστάθμιση κινδύνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Πατράου Νέβες Γιάρ και μετά η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει ίσως ε, να προχωρήσουμε ε, με δύο διαφορετικούς τρόπους ε, και τελώς κάποιος ε, που προέρχεται από τη Γερμανία σε σοσιαλιστικό καθεστώς. Πολλά από αυτά που άκουσα μου φάνηκαν γνωστά. Παλαιότερα στη σοσιαλιστική Γερμανία είχαμε σταθερές τιμές στη Γεωργία, δεν είχαμε κερδοσκοπία. Η αξία της γης, της γεωργικής γης ήταν μηδενική, κανείς δεν μπορούσε να αγοράσει αξία. Δεν είχαμε βέβαια χρεοκοπίες ε, Παρ' όλα αυτά κάποια στιγμή το σύστημα δεν ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθεί διότι δεν έλειφθη υπόψη η επιχειρηματικότητα και διότι δεν υπήρξαν καινοτομίε. Άρα δηλαδή το πρώτο θέλω οπωσδήποτε να το ε, υποστηρίξω ότι πρέπει να απευθυνθούμε στον Γεωργό με την ιδιότητά του του επιχειρηματία. Να τον ενθαρρύνουμε στην επιχειρηματικότητά του. Βεβαίω και πρέπει να λειτουργεί η αγορά και εδώ ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Νταντάν, δηλαδή ποιο θα δώσει τι απαραίτητε πληροφορίες στους γεωργούς. Ίσως εδώ οι γεωργικοί συνεταιρισμοί να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό. Η γεωργία ε, προφανώς έχει και το καθήκον της, ε, του εφοδιασμού με τρόφιμα. Εδώ μπορούμε να καταφύγουμε σε κάτι που είπε ο Λένιν. Ο Λένιν είχε ήδη πει τότε το σιτάρι είναι όπλο. Ο Λένιν δηλαδή το είχε ήδη τότε συλλάβει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει επαρκής εφοδιασμός τροφίμων για τους πολίτες. Άρα δηλαδή με τη γεωργία ασκούμε και πολιτική ασφαλείας. Και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς. Εδώ, τίθεται το ερώτημα της επιστροφής των εξαγωγών. Ε, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο πράγματι. Οι ποσοστώσεις να υπάρχουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι αν είμαστε ειλικρινείς με τις ποσοστώσεις γάλακτος αποτύχαμε. Διότι απλούστατα η πολιτική δεν ήταν σε θέση να προσαρμόσει την ποσόστοση στις ανάγκες της αγοράς. Επιτρέψαμε υπερβολικές πεσότητες και παρόλα αυτά οι ε, τιμές έπεσαν. Ε, γι' αυτό λοιπόν τίτε το εξή ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να επιτύχουμε ισορροπία αφενός γεωργική επιχειρηματικότητα, και καινοτόμος γεωργία, από την άλλη όμως να μην παραμελούμε και το στοιχείο της πολιτικής ασφαλείας που σας εξήγησα. Οφείλουμε την ε, μάλλον η γεωργική μας πολιτική πρέπει να είναι σε θέση να θρέψει τους 500 ε, εκατομμύρια κατοίκους, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην είμαστε εξαρτώμενοι από άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γιά. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης ε, ε, και για αυτά που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από πλευρά οικονομική και γεωργική πλευρά. Ε, πολύ χρήσιμα αυτά που είπε και ο κύριο Γιάρ με βάση την εμπειρία του. Δύο παρατηρήσει έχω να κάνω. Η πρώτη μου ερώτηση έχει σχέση με τι ε, διακλαδικέ οργανώσει, οργανώσει παραγωγών για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ε, περισσότερες πληροφορίες για το πού λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το μοντέλο. Νομίζω στη Γαλλία είναι, έχει ριζώσει περισσότερο και ποιες είναι οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πολυκλαδικές οργανώσεις και οργανώσεις παραγωγών λειτουργούν αποτελεσματικά. Τα σχόλια που έχω να κάνω έχουν σχέση με την παραγωγή ε, σχετικά με τις τιμές, ε, με τη διατροφική αλυσίδα, το εισόδημα, τη μεταφορά προϊόντων δεν ξέρω αν θα πρέπει να μετρήσουμε το εισόδημα από τη Γεωργία. Γιατί κοιτάξτε, το εισόδημα μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, τα χρήματα που κερδίζουν οι άνθρωποι από τη Γεωργία. Και οι τάσεις που επικρατούν σχετικά με αυτό. Είναι υποκρισία να λέμε ότι αν ένα νοικοκυριό έχει εισόδημα από άλλη πηγή, προστίθεται αυτό στο γεωργικό εισόδημα. Δεν είναι εισόδημα από τη Γεωργία και πρέπει να μετριέται ξεχωριστά. Η δεύτερη μου έχει σχέση με την αξία της γης. Πραγματικά εκπλήσωμαι που όλοι σας εκπλήσεστε ε, ότι αυξάνεται η αξία της γης ακόμα και αν πέφτει η γεωργία. Μα η, η υγεία είναι οικονομικό αγαθό ε, η ποιότητά της ε, πέφτει, γι' αυτό λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο να αυξηθεί η τιμή της. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Και τέλος θέλω να πω, οι πολύ πλούσιοι οι οποίοι αποκτούν ε, χρήματα από άλλους τομείς χάνουν χρήματα από τη γεωργία. Και άκουσα κάτι τέτοιο αλλά δεν το κατάλαβα και δεν το καταλαβαίνω ποτέ όταν τα ακούω. Θα ήθελα λοιπόν οι τιμές ε, της έγκυας ιδιοκτησίας ε, να παραμείνουν σταθερές, ε, και ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το πετύχει αυτό με τα βιοκάψιμα. Δηλαδή η γη πρέπει να παράγει τρόφιμα, καύσιμα, ίνες, ε, δημόσια αγαθά. Άρα δηλαδή η πίεση στη γη θα αυξηθεί, θα κληθεί η γη να προσφέρει όλα αυτά τα προϊόντα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έλλειψη αυτού του προϊόντος ε, της γης. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ε, τελείωσε λοιπόν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και στο ε, σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές μας και θα ήθελα... Α, θέλουν να απαντήσουν. Μισό λεπτό. Έχει το λόγο ο εισηγητής για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ο κύριος Γκοέν, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να απαντήσω. Θα προσπαθήσω να είμαι ακριβής. Για την πρώτη παρέμβαση υπόθηκε ότι οι αγορές θα μπορούσαν να βοηθήσουν για τη διαχείριση του κινδύνου. Ναι, αλλά δεν ισχύει για όλες τις παραγωγές. Δεν μπορεί να φανταστεί δηλαδή κανείς ε, ότι θα μπορούσε να ισχύει αυτό για την ντομάτα και το καρότο για παράδειγμα. Όσον αφορά τους συνεταιρισμούς που είπατε εσείς ότι είπα ότι είναι πολύ ισχυροί. Ε, ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, ε, αυτό εκεί θα έπρεπε να είναι η ισχύ στους συνεταιρισμούς. Όσον αφορά τώρα το ΠΟΕ και την αποσταθεροποίηση των παγκοσμίων αγορών. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά που λέει ο ΠΟΕ. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τις παγκόσμιες αγορές. Και όταν μιλάμε για παράδειγμα για μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ασφάλεια των αγορών, είναι σαν το σύστημα marketing loan ε, του 1996 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, βάσει της ιστορίας ε, δηλαδή αναθεωρούσαν τις τιμές. Δεν μιλάω τώρα για το, για το παρόν, μιλάω για την παρελθούσα κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, όσον αφορά την ποσοτικοποίηση που έγινε στην αξιολόγηση αντικτύπου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια απόδοση από τις επενδύσεις για τις οποίες μιλήσατε, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μποβέ για τους ε, ε γεωργούς. Η αναδιάρθρωση ήταν ε, ήδη ένα πολύ καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση το γεγονός ότι καταργήθηκαν κάποιες ποσοστώσεις ε, θα δημιουργήσει ενδεχομένως 2 ε, ε, με 5% μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά όχι παραπάνω. Κοιτάξτε, πρέπει να σας ομολογήσω ότι είχα πάρα πολλές συζητήσεις με τους ανθρώπους του κλάδου στη Γαλλία για όλο αυτό το θέμα των ποσοστώσεων γάλακτος ή ποσοστώσεις γάλακτος. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό είναι επικερδής ε, μόνο για ε, όσους βρίσκονται επί τόπου εκείνη τη στιγμή. Μετά όσοι ε, έρχονται εκ των υστέρων στον κλάδο δεν τους βοηθάει καθόλου. Βοηθά μόνο εκείνους που είναι στο επάγγελμα όταν δημιουργούνται. Από εκεί και πέρα πρέπει κανείς να πληρώσει ένα τίμημα και κανείς δεν συμφωνεί, τουλάχιστον από τους ανθρώπους του κλάδου με τους, του κλάδου με τους οποίους εγώ ήρθα σε επαφή, δεν μπορώ να καταλάβω, κανένας δεν μπορεί να αποφασίσει το επίπεδο. 5-10%. Όλοι πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν την προσπάθεια και όχι ο ίδιος ο γεργός στη δική του γεωργική εκμετάλλευση ή στη δική του χώρα. Όσον αφορά τις άμεσες ε, ε, ενισχύσεις και κατά πόσο θα μπορούσαν να έχουν ε, αρνητικό αντίκτυπο στο γεωργικό εισόδημα. Πάρα πολλέ μελέτε υπάρχουν που συμπεραίνουν ότι οι άμεσε ενισχύσει, όχι την πρώτη χρονιά, αλλά σε 5-10 χρόνια, ανάλογα με την έγκυο ιδιοκτησία τη κάθε χώρα, τελικά φτάνουν στου γεωκτήμονε και μόνο και δεν φτάνουν στους ε, ε, γεωργού. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί ε, ιδιοκτήτε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, είναι 80% στο σύστημα, στο ε, Οπότε είναι γεγονός ε, ότι αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι την ύφη πρέπει να την πληρώσει τελικά ο Γεωργός ο ίδιος. Και ποιο, ε, και ποιο είναι το αποτέλεσμα Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υποστηρίξουμε τους οικονομικούς φορείς που παράγουν αγαθά. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ όλο και περισσότερο να ε, ε, εισαγάγουμε όρους για τις άμεσες ενισχύσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να επιμένουμε πάρα πολύ ε, στην ε, ε, διαβάθμιση, γιατί νομίζω ότι είναι διαφορετικό πράγμα η υποστήριξη η ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και διαφορετικό πράγμα αυτό που προτείνω εγώ. Μπορούμε να μειώσουμε τις διαρροές. Από τη στιγμή που υπάρχει μια πολιτική υπάρχουν διαρροές. Από τη στιγμή που δίνουμε ένα ποσό στο, στο γεωργό, πάντοτε θα υπάρξουν κάποιες διαρροές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς είναι δυνατόν να τον ενισχύσουμε περισσότερο για να μπορέσει να προβεί στην παραγωγή των αγαθών που χρειάζονται δεν ε, υπάρχει ας πούμε το θέμα του σεβασμού των περιβαλλοντικών ε, προδιαγραφών. Υπάρχει για παράδειγμα ένα πρόγραμμα που επιβάλλει στους γεωργούς της Γαλλίας ε, ε, μείωση ε, δίνει δυνατότητα μείωση τιμών 50% για τα αντιβιωτικά, για παράδειγμα, σε περίπτωση κάποιας ασθένειας, αν πληρούν κάποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Όλο και περισσότερο πρέπει να στο, στοχεύουμε το ενεργό γεωργικό πληθυσμό και δεν πρέπει να λέμε αν ναι, θα δούμε μετά στη συνέχεια αν θα έχουμε τα χρήματα να, να βοηθήσουμε ή όχι». Όσον αφορά τώρα τους επαγγελματίες, ε, ε, υπήρχε μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, ε, κυρίως για, τα, για τον τομέα των φρούτων. Η εσωτερική αγορά ε, μπορεί να αποδώσει σε βάθος χρόνου ενός-δύο ετών, ενδεχομένως ο κύριος Μποβένα το ξέχασε αυτό, δεν χρησιμοποιούν την εσωτερική αγορά υποχρεωτικά όλοι οι γεωργοί ή μόνο οι γεωργοί. Υπάρχουν και εκτινοτρόφοι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον, κάποιο, κάποια ένδειξη στην οποία να μπορούμε να βασιστούμε. Απλώς αυτό που είπα είναι ότι αν βασιστούμε στον κλάδο υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Και για να μην μακρηγορώ, με ρωτήσατε για παράδειγμα για την κερδοσκοπία. Πρέπει να επιβεβαιώνουμε ότι στις εσωτερικές αγορές δεν υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Σε αυτό συμφωνώ απολύτω. Δεν είμαστε και πρωτοστάτε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι Ηνωμένε Πολιτείε τα πάνε πολύ καλύτερα. Ελπίζουμε ότι θα προωθήσουμε, αλλά, θα προοδεύσουμε, αλλά δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι για την ώρα τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα τους μικρούς ε, γεωργούς, με, ρωτούσατε, ρωτήσατε αν κάναμε μεγαλύτερη διαβάθμιση, ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εγώ συμφωνώ να στοχεύσουμε περισσότερο στους μικρότερους γεωργούς, σε πάση περιπτώσει στο ενεργό δυναμικό της γεωργίας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω, χωρίς να είμαι βέβαιος ότι έχω καλύψει όλες τις ερωτήσεις, εγώ θα πρότεινα τουλάχιστον να λάβουμε υπόψη δύο ιδιαιτερότητε τη γεωργία. Πρώτον, δεν μπορεί κανεί να απαγορεύσει σε ένα κράτο μέλο να παρέμβει όταν πιστεύει ότι υπάρχει λόγο να το κάνει. Το 2008, για παράδειγμα, υπήρξαν ε, τεράστιε εξεργέρχε λόγω τη πείνα που δεν είχαν να κάνουν απαραίτητο με την επισητιστική ασφάλεια. Υπήρχαν προβλήματα με τι ε, τιμέ ενέργεια, για παράδειγμα. Ε, όταν όμως παίρνουμε μια, ε, ε, ένα καρβέλι ψωμί και βγαίνουμε στους δρόμους, από απόψε ως δημοσίευσης ε, είναι πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα που στέλνουμε. Αυτό, που βασίζω, αυτό που, που, στο οποίο βασίζονται οι άνθρωποι αυτοί είναι κυρίως ο φόβος που μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια εικόνα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αν ο καθένας ασχολείται μόνο με τη δική του αγορά, ε, μπορεί να δημιουργήσει στρέβλωση στην παγκόσμια αγορά και πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους ιστορίες. Ε, όλοι φοβούνται μήπως η Αργεντινή, μήπως η Ρωσία ε, κλείσει τα σύνορά της στις εισαγωγές. Ναι, αλλά πρέπει όλα αυτά να το τοποθετούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη ε, ε, ιδιαιτερότητα της γεωργίας και η δεύτερη είναι η ίδια η γη. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι η τιμή της γης ε, είναι υψηλή ή χαμηλή. Είπα απλώς ότι όταν αυξάνεται η χαμηλη ειπα απλω υπάρχουν οικονομικοί φορείς που το πληρώνουν αυτό το τίμημα. Διαφορετικά δεν θα επληρώναν ακριβά την τιμή της γης. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα επίσης της γεωργίας και είναι και ένας δείκτης που πρέπει να τον παρακολουθούμε είναι πιο ενδιαφέρον όταν βασιζόμαστε ε, στις πληρωμές των γεωργών ε, παρά στις δηλώσεις τους. Γιατί οι δηλώσεις ε, πάντα αρνητικέ θα είναι. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτές. Μετά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να κάλυψα τα ερωτήματά σας κατά το μέγιστο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό το θέμα. Ευχαριστούμε τον εμπειρογνώμονα μας και θα επανέλθουμε φυσικά σε αυτό το θέμα της διαχείρισης κινδύνων θα αποτελέσει αντικείμενο γενικότερης σκέψης και θα εμπλουτίσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κάπουλα Σάντος, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στα σχόλιά της μία απάντηση στο αίτημά μας ε, για πληροφορίες στις διαφόρες, για τις διάφορες προσωμιώσεις που έγιναν στα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια της χαρτογράφησης των ε, μειονεκτουσών περιοχών αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο παρέμβασης και στην Ολομέλεια από πλευράς ε, ε, βουλευτών. Γι' αυτό να το λάβετε υπόψη. Ο Λουίς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε αυτή την δυνατότητα, λοιπόν, να ακούσουμε τους συναδέλφους ε, για αυτή την πρόταση κανονισμού θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Επιτροπή γιατί ως προς το σύνολο των κανονισμών ε, είναι ο καλύτερος. Είτε πρόκειται για οργανώσεις, αγροτικές οργανώσεις ή εθνικές κυβερνήσεις. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι στον απογραφικό κατάλογο αναφέρονται οι προτεραιότητες που υποστηρίζουμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ως προς τις βασικές προτάσεις για την μελλοντική εκλογιμότητα, επιλεξιμότητα με συγχωρείτε, μιλάμε για τα κίνητρα για συστήματα ποιότητας, επιδοτήσεις ως προς τα ασφαλιστικά καθεστώτα για την εμπορία και μεταποίηση, επίσης ανταπόκριση στις φυσικές καταστροφές και εδώ θα πρέπει να διευρύνουμε το πλαίσιο δράσης για να συμπεριλάβουμε και την ξηρασία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε δηλαδή και σε άλλες καταστροφές ε, γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη επαρκώς η ξηρασία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση οικονομικής ε, βάσης και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τους νέους γεωργούς. Υπάρχουν πολλά χάσματα και δεν δίνονται κίνητρα για την προσβασιμότητα στη γη και δυστυχώς δεν συμμετέχουν νέοι στην επίμορτο αγροληψία. Επίσης θα πρέπει να τονώσουμε τις ε, υποδομές και τις βασικές υπηρεσίες για τις κομοπόλεις, για τα δάση και να υποστηρίξουμε τις ε, οργανώσεις παραγωγών. Πέρα όμως από τις ε, χρηματοοικονομικές, από τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς, θα πρέπει να μας απασχολήσει η ε, επιλεξιμότητα περιφερειών. Επίσης, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ε, επηρεάσουμε αυτά τα μέτρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει στο greening, στο πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα να ληφθούν υπόψη και τα ε, αγροτοπεριβαλλοντικά προϊόντα, να εφαρμοστεί λοιπόν το πρασίνισμα και να μπορέσουν να ισχύσουν και οι δύο αυτοί πυλώνες. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την Natura 2000 στην οδηγία για τον υδροφόρο ορίζοντα και όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή για τα κράτη-μέλη, να δούμε ποιες είναι οι εδαφικές επιπτώσεις κατά την οριοθέτηση αυτών των περιφερειών και ε, ε, μας ενδιαφέρει και η ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου και τα μέτρα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο Επίσης, οι επιδοτήσεις για την καινοτομία και την ενδυνάμωση των αγορών. Γι' αυτό θα πρέπει μέσα στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα να υποστηρίξουμε τους μικρούς αγρότες, να διασφαλίσουμε τη συγκομιδή, να ε, αποτρέψουμε ασθένειες στην πανίδα και την χλωρίδα και θα πρέπει αυτό το περιεχόμενο να αποσαφινιστεί επαρκώς έτσι ώστε να είμαστε αποδοτικοί. Είμαστε υπέρ του leader, μιλάμε για χρηματοδότηση που ανέρχεται στο 5% και δεν ξέρω κατά πόσο το leader στο μέλλον θα μπορούσε να υποστηρίξει ε, δάφη που δεν έχουν αγροτικό χαρακτήρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Λίντερ τάσεται υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης και θα πρέπει να δούμε τι άλλα μέσα έχουμε για αυτό το σκοπό και τέλος μας ενδιαφέρει η καινοτομία θα πρέπει να δώσουμε οικονομικά κίνητρα στην καινοτομία και η Επιτροπή μιλά για χρηματοοικονομική πρικοδότηση δυνάμει του κάπινγκ του πρώτου πυλώνα, δηλαδή των οροφών, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κοινοτική χρηματοδότηση 100%. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να, το, να τονίσουμε. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα προς απόφαση. Ως προς την κατανομή του προϋπολογισμού του δεύτερου πυλώνα, γιατί η Επιτροπή στον πρώτο πυλώνα προτείνει στο δεύτερο παράρτημα κατανομή ανακράτος μέλος, αλλά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποθεματικό και ποια κριτήρια θα ακολουθήσουμε για την ε, κρατική κατανομή. Δεν μπορούμε παρά να προτείνουμε κάτι το συγκεκριμένο. Αυτό αφορά την Επιτροπή διότι το θέμα είναι αμφίσιμο δημοσιονομικά. Θα πρέπει όμως ε, το Κοινοβούλιο να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα άλλο θεσμικό όργανο για να αποφασίσει μεμονωμένα επί του θέματος. Ε, θα ήθελα λοιπόν να φτάσουμε σε μία συνενετική ε, φόρμουλα για το δεύτερο πυλώνα. Και επίσης την συμπερίληψη του πρασινίσματος στον τομέα των αγροτικό και περιβαλλοντικό για να λάβουμε υπόψη το greening στον πρώτο πυλώνα. Υπάρχουν και άλλες παραλήψεις, δηλαδή ως προς την πάυση δραστηριοτήτων η Επιτροπή ήρε αυτή τη ρήτρα. Γιατί αν υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα και εάν υπάρχει γύρανση του πληθυσμού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί διότι η ενεργός ζωή παρατείνεται και γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε μία πρόταση επί του θέματος. Ως προς την συγχρηματοδότηση θα πρέπει να ορίσουμε τους δείκτες συγχρηματοδότησης και να δούμε τι προτείνει η Επιτροπή, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και να υπάρχει ιδιωτική συγχρηματοδότηση στο αγροτικό περιβάλλον. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες σε ορισμένα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να τις αποτρέψουμε. ιδιαίτερα όταν υπάρχει ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η προσέγγιση μου και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να φτάσουμε σε συνενέσεις εδώ, καλύτερα παρά στις άμεσες πληρωμές όπου υπάρχουν μεγαλύτερες αμφισημίες. Και είμαι στη διάθεσή σας για να δεχτώ τη θέση των σκιωδών και των συναδέλφων και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει τους εισηγητές για να έχουμε μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι του Συμβουλίου. Έχει μεγάλη σημασία η μεγάλη μας διαπραγματευτική δύναμη και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε Λουίς. Ας ξεκινήσει λοιπόν ε, η συζήτηση με την Elizabeth Κόστιντζερ και μετά ο Αντρός Πόλσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή, τον Λουίς Κάπολα Σάντος, για την εισαγωγή του στο θέμα αυτό που είναι η γεωργική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Εγώ ε, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η συγητής, που είπε ότι η αγροτική ανάπτυξη αντιμετωπίζεται ως κάτι το εύκολο ε, στα πακέτα που παρουσιάζει η Κομισιόν. Όμως ε, παρόλα αυτά δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που είναι πολύ δύσκολες. Θέλω να πω το εξής οι ε, εταιρικέ συμβάσεις που προτείνονται τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφήγησαν, δεν αναφέρθηκαν, όμως θα ήθελα να επισημάνω το θέμα αυτό και αρμόδια ε, δεν θα είναι μόνο η Επιτροπή Γεωργίας αλλά και η Επιτροπή των Περιφερειών. Οφείλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα ψηφοφορίας γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να περιοριστεί η επιρροή της Γεωργίας στα προγράμματα ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε στον ε, αγροτικό τομέα. Επιπλέον σε αυτόν τον τομέα φοβάμαι ότι είναι δυνατόν να αυξηθεί ε, κατά πολύ το διοικητικό άχθος ε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Να σκεφτούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά στα παραρτήματα Προπολογισμού που προτείνει ο εισηγητής στον τομέα της γεωργίας, εκεί θα ήμουν πολύ προσεκτική. Στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών είχαμε πολλές και ζωντανές συζητήσεις όσον αφορά τον επιμερισμό των κονδυλίων. Και παρότι είναι σημαντικό να βλέπει κανείς από κοινού τους δύο πυλώνες της ε, γεωργικής πολιτικής, παρόλα αυτά ο πυλώνας υπαριθμών 2, η γεωργική ανάπτυξη, έχει τελείως διαφορετικά κριτήρια από τον πρώτο. Δηλαδή δεν στηρίζονται τα μέτρα της αγοράς, αλλά αυτό που παίζει ρόλο είναι οι επιπρόσθετες υπηρεσίες ε, που προσφέρει ο Γεωργός. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι πολιετής και συγχρηματοδοτούνται. Άρα δηλαδή, ε, ναι, βλέπει κανείς αυτούς τους δύο πυλώνες από κοινού, αλλά παρόλα αυτά διαφοροποιημένα. Και να πω και κάτι σχετικά με τις ενισχύσεις ε, στο δεύτερο πυλώνα. Παραδείγματο χάρη στην πρόταση της ε, Επιτροπής δεν γίνεται λόγος, δεν αναφέρεται ο ορισμός του ενεργού αγρότη. Όμως ο όρος αυτός ενεργός αγρότης παίζει μεγάλο ρόλο στο δεύτερο πυλώνα. Δηλαδή ο ενεργός αγρότης ε, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα πρόγραμμα παρότι ενδεχομένως ε, να μην έχει ο ίδιος ε, αρμοδιότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Επίσης, οι μικροί γεωργοί αυτοί πρέπει να εξαιρούνται από τις διατάξεις της πολλαπλής συμμόρφωσης στον πρώτο πυλώνα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλους ε, τους ε, παράγοντες ε, και όλους εμπορευόμενους να τους βλέπουμε μέσα σε έναν συνεταιρισμό και να στηρίζονται στο πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης. Αυτό αναφέρεται ε, παλαιότερα, αλλά όχι σε αυτή την πρόταση που έχει κατατεθεί. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο κατά την άποψή μου που έχει σχέση με την γεωργική ανάπτυξη είναι τα γεωργικά και τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Και εδώ συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του εισηγητή ότι θα πρέπει τους δύο πυλώνες να τους εξετάζει κανείς από κοινού. Και οφείλουμε να κάνουμε μια σε βάθος συζήτηση για τα 25% ε, δαπάνω πάνη του 25% για το περιβάλλον, αυτά ε, αναφέρονται μόνο στο σκεπτικό, πουθενά άλλου. Και θεωρώ ότι τα γεωργικά και τα περιβαλλοντικά προγράμματα πρέπει να είναι πολύ σωστά πρικοδοτημένα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα ωφελήσει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση του εισηγητή ότι στο πλαίσιο του πρασινίσματος οι εκμεταλλεύσεις ε, ε, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν με πολύ καλά προγράμματα βέβαια δεν είναι απαραίτητο να πληρούν τις προδιαγραφές του πεσενίσματος στον πρώτο πυλώνα. Και θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό τον τομέα και η πρόταση της Κομισιόν ως έχει διαμορφωθεί τώρα η πρόταση αυτή είναι οπισθοχώρηση για τα κράτη αυτά όχι μόνο οικονομικής φύσεως αλλά και όσον αφορά την αποδοχή των προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι ως εκπρόσωποι των γεωργών και των ψηφοφόρων μας ε, καλούμεθα να είμαστε ε, πολύ ε, προσεκτικοί γιατί σε τελική ανάλυση εδώ πρόκειται για την αποδοχή της πολιτικής μας. Όσον αφορά τώρα ε, τις ε, μειονεκτούσες περιοχές, εκεί υπάρχουν κατά την άποψή μου ορισμένα ε, κρίσιμα θέματα. Θα υπάρξουν αλλαγές στα λογιστικά συστήματα. Ιδιαίτερα προβληματικό είναι αυτό που αναφέρεται σχετικά με το ύψος του, της πρημοδότησης 300 ευρώ ανά εκτάριο κατά το μέγιστον. Αυτό διαφοροποιείται από το τελευταίο πρόγραμμα της γεωργικής ανάπτυξης. Και εδώ έχουμε πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές προφανώς στις μειονεκτούσες περιοχές, στις ορεινές περιοχές όπου κάποιες εκμεταλλεύσεις είναι εκτός αυτού του ανώτατου ορίου αλλά και διότι ασχολούνται ε, ενεργά με τη γεωργία και βρίσκονται σε απομακρυσμένη και μειονεκτούσα περιοχή. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι να παραμείνει ενεργή γεωργία στις μειονεκτούσες ε, περιοχές. Όσον αφορά την ε, επαναξιολόγηση των υπόλοιπων μειονεκτουσών περιοχών, ο πρόεδρος το είπε στην αρχή, αναφέρθηκε στην συζήτησή μας με το Συμβούλιο, και επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναντάτες και τις πολιτικές ομάδες που ε, το ερώτημα αυτό στηρίχθηκε ανεπιθύλακτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να καλέσουμε το Συμβούλιο να διευκρινίσει το θέμα αυτό. Ε, δεν είναι σωστό να μην προβούμε σε διαφοροποίηση και θα συνέβαινε κάτι τέτοιο εάν δεν τοποθετούμε πάνω σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν είναι ικανοποιητική λύση αυτών των, της αξιολόγησης των οκτώ βιοφυσικών ε, κριτηρίων. Σε ορισμένα κράτη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το Συμβούλιο και οι Κομισιόν καλούνται να διευκνήσουν περαιτέρω το θέμα αυτό. Όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Ε, εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα γιατί οι πολιτικές μας ομάδες ασχολήθηκαν σε βάθος με το θέμα αυτό. Δηλαδή κατά πόσον η διαχείριση κινδύνων είναι λογικό να υπάρχει στον δεύτερο πυλώνα ή όχι. Αυτή τη διαχείριση κινδύνων την έχουμε ήδη μέσω του άρθρου 68 στον πρώτο πυλώνα. Αυτό κατά το παρελθόν βέβαια. Η διαχείριση κινδύνων είναι ένα κλασικό εργαλείο διαχείρισης αγοράς και άρα ο δεύτερος πυλώνας δεν ενδείκνυται και νομίζω ότι πρέπει να εξτάσουμε ε, επί της ουσίας το θέμα αυτό. Όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση και εκεί ισχύει το ίδιο. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εξαιρούμε τομείς ε, και προβλέπουμε μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση, αυτό όμω σημαίνει αυτόματα ιεράρχηση. Ε, δηλαδή ε, σε κάποιους τομεί περισσότερα χρήματα, σε άλλου λιγότερα. Ε, το θέμα λοιπόν της συγχρηματοδότησης πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ για να έχουμε αίσιο τέλος. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στα δασοκομικά μέτρα που αναφέρονται στον δεύτερο πυλώνα. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικό το ότι το θέμα της ανταγωνιστικότητας εξαιρείται από τη δασοπονία και δασοκομεία. Εγώ ε, θεωρώ ότι πρέπει να εξετάζεται, κυρίως όταν πρόκειται για καταβολή ενισχύσεων. Και ιδιαίτερα προβληματική βρίσκω την πρόταση ότι οι δασοκομικές εκτάσεις ε, πρέπει να υποβάλουν προγράμματα. Αυτό όμως για μικρές εκμεταλλεύσεις ε, δημιουργεί ε, περισσότερο αύξηση του κόστους και δεν αιτιολογείται το κόστος αυτός με ανάλυση κόστους ωφέλους. Ε, στον τομέα λοιπόν της δασοκομείας πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Οι προτάσεις της Επιτροπής για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τη βιομάζα στον τομέα της δασοκομείας, αυτή η πρόταση είναι καλή. Γιατί θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι σημαντικό και σε σχέση με τους στόχους του 2020. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον εισηγητή ε, για αυτή την ε, πρώτη παρουσίαση της έκθεσής του. Ε, προσβλέπω στην συνεργασία κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής. Ο Αντιπρόεδρος κ. Πόλτσον έχει το λόγο. Ή Αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε. Ett bra början Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια πολύ καλή αρχή ε, και θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξής, ε, ότι η πόλη και η πετρός είναι ένα ενιαίο σύνολο. Είναι αδύνατον να ε, σκεφτόμαστε το μέλλον της Ευρώπης χωρίς να έχουμε κατά νου ζώντα χωριά με ζωή, γεωργία και δασοκομεία με ζωή. Η εύρυθμα λειτουργούσα γεωργία είναι ανεξάρτητη από το ευρύτερο περιβάλλον, ανεξάρτητη από τους καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μία διασύνδεση ανάμεσα σε όλα αυτά τα θέματα και θέλω να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις όσον αφορά την ιεράρχηση και συγκεκριμένα το άρθρο υπαριθμών 5. Θα μιλήσω καταρχήν μόνο για τη γεωργία και όχι για υπόλοιπα θέματα που αφορούν τα χωριά και την Ήπετρο. Αναφέρομαι σε εγκαταστάσεις υδροδότησης. Ε, στο θέμα αυτό ε, θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Κάτι που να είναι σημαντικό για το σύνολο του συστήματος και όχι για μεμονωμένους γεωργούς. Οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε τα συστήματα της συντροδότησης, κυρίως Αναφέρεται εδώ αν είναι δυνατόν να υπάρξει εξοικονόμηση τη τάξη του 25%. Αυτό όμω είναι λάθο. Αλλιώ έπρεπε να διατυπωθεί η πρόταση. Να γίνεται λόγο για αποτελεσματικό σύστημα υδροδότηση που οδηγεί σε εξοικονόμηση και επίση σε καλύτερη χρήση των, ε, του τμήματος της ποσότητας εκείνης ε, των υδάτων που χάνονται στον αέρα. Να μπορούν αυτά, παραδείγματος χάρη, να, τα, τα νερά να ψεκάζονται πίσω για την καλλιέργεια της ντομάτας. Εάν λοιπόν ε, έχουμε καλές εγκαταστάσεις υδροδότησης, παραδείγματος χάρη στη Μεσόγειο, Αυτό επιτρέπει ε, καλύτερη πρόσβαση ε, και στο βορρά. Έχουμε δηλαδή ε, ποιοτικά, περισσότερο ποιοτικά οπωροκυπευτικά, κυρίως κατά την περίοδο όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς. Και εάν υπάρχει λοιπόν ευφυής παραγωγή, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση για το σύνολο της Ευρώπης. Αυτά για το νερό. Όσον αφορά τώρα τα βιοκαύσιμα, πρέπει να σας πω, χαίρομαι ιδιαίτερα που στο έγγραφο της Κομισιόν αναφέρεται ότι ε, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προϊόντα τα οποία ναι είναι αποδομήσιμα αλλά δεν είναι βρόσιμα. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα στην αξία της γης. Κατά πόσον η αξία της γης είναι συνδεμένη με τις τιμές ενέργειας στην παγκόσμια αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτάρκεια στη γεωργία μας, έτσι ώστε οι γεωργοί να απελευθερωθούν από, τις, από την επιρροή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Αυτά είχα να σας πω. Και κάτι άλλο που έχει σχέση με το δεύτερο πυλώνα. Ο πρώτος πυλώνας, στον πρώτο πυλώνα γίνεται λόγος για την αποκαλούμενη οικολογικοποίηση της παραγωγής, δηλαδή γίνεται λόγος για το ότι πρέπει να καλλιεργηθούν διάφορα φυτά, ε, να χρησιμοποιηθούν οι εκτάσεις που υπάρχουν. Γίνεται όμως εκεί λόγος και για τις μειονεκτούσες ε, περιοχές. Γίνεται λόγος, ας πούμε, και για την γεωργία στην Αρκτική. Αυτή η παραγωγή είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό στις ε, περιθωριακές ε, περιοχές, στις άκρως απομακρυσμένες, να έχουμε γεωργία ζωντανή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν προβλήθηκε αρκετά. Εγώ θα ήθελα να αναφέρεται ως ε, προτεραιότητα. Και επίσης θα ήθελα να υπάρχει και διασύνδεση με την όλη προβληματική που έχει σχέση με θέματα υγείας. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την One Health Strategy, όπως λέγεται αυτή τη στρατηγική υγείας, που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την ζωική παραγωγή. Μην ξεχνάτε τους κλοβούς, ε, την ε, παραγωγή πουλερικών σε και νομίζω ότι και αργότερα θα ασχοληθούμε με την ε, καλή διαβίωση των ζώων, κυρίως στην εκτροφή των χείρων. Όσον αφορά τι επενδύσεις, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα επένδυσης σε καλύτερα συστήματα εκτροφής. Συστήματα καλύτερα για τα ζώα αλλά και για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα συνδυασμών έτσι ώστε να έχουμε ένα σύνολο με πολλές αποχρώσεις. Πολύ συχνά οι προτάσεις που υποβάλλονται είναι κατατριμμένες, περιλαμβάνουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να έχουμε μπροστά μας ένα σύνολο, ένα σφαιρικό πρόγραμμα και ε, να γνωρίζαμε το σύνολο του μοσαϊκού. Βασικά σημεία θα πρέπει να είναι η υδροδότηση, η ενέργεια και η κτηνοτροφία. Μία κτηνοτροφία φιλική προς τα ζώα. Ευχαριστούμε Πρίτα Ρέιμερς και Μάρτιν Όσλικ. Ε, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που με ενδιαφέρει, στη συγχρηματοδότηση. Η συγχρηματοδότηση μας προκαλεί προβλήματα. Με την έννοια βλέπουμε όλο και περισσότερες περιοχές και κράτη τα οποία έχουν πρόβλημα να βρουν τα κονδύλια για τη συγχρηματοδότηση. Άρα δηλαδή πρέπει να βρούμε κάποια λύση για το πώς ε, ε, θα διαμορφωθούν στο μέλλον τα προγράμματα έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ε, λογικής και εύρυθμης ε, ροής των κονδυλίων. Γιατί ε, τα κράτη χρειάζονται τα κονδύλια για να αναπτύξουν τις περιοχές τους. Γι' αυτό λοιπόν εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακριβώς όπως και στο Περιφερειακό Ταμείο, το Ταμείο Αλίας, ε, το Κοινωνικό Ταμείο, ταμεία με τα οποία ε, καλούμεθα να συνεργαστούμε, με αυτά να έχουμε μια καλύτερη δυνατότητα συγχρηματοδότησης έτσι ώστε όπως σας είπα να ρέουν τα κονδύλια διότι χρειαζόμαστε μια γεωργία η οποία θα εντάσσεται στην ευρύτερη οικονομία της ε, Υπέτρου ε, Ταμείο Γεωργίας ε, και, Γεωργικό, και Περιφερειακό Ταμείο και Γεωργικό Ταμείο πρέπει να βελτιωθούν να δουν που υπάρχουν επικαλύψεις πώς είναι δυνατόν να επιθε... αποφευθούν οι επικαλύψεις διότι αν δεν ενισχύσουμε τη γεωργία και αν δεν ε, πετύχουμε την ε, σταθερότητά της, ε, θα έχουμε απερίμωση. Οι νέοι θα μετακινηθούν περισσότερο προς τις πόλεις. Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε μεγαλύτερη αστιφιλία στην Ευρώπη και ελοχεύει ο κίνδυνος τα σχολεία πλέον είναι πολύ ακριβά για να παραμείνουν στην Ήπετρο ή και οι ε, παροχές υπηρεσιών υγείας και αυτό πολύ δαπανηρό ή αν θέλετε οι ε, δυνατότητες για τα νοικοκυριά να ε, αποκτήσουν τα πρώτα αγαθά η μέρημνα για τους ηλικιωμένους. Όλα αυτά γίνονται ε, πολύ δαπανηρά και αυτές ε, είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη σταθερότητα της ε, γεωργίας. Και αυτό λοιπόν όλα αυτά σημαίνουν ότι τα κονδύλια πρέπει όπως σας είπα να εκταμιεύονται προς τη γεωργία. Και κάτι άλλο. Κατά την τελευταία περίοδο διαπιστώσαμε ότι στην αρχή υπήρχε μία στασιμότητα ε, μέχρι να αρχίσουν να εκταμιευτούν, να αρχίσουν να εκταμιεύουν τα κονδύλια προς τη Γεωργία. Και τώρα που βρισκόμαστε ε, στο, στην τελευταία φάση ε, μεταρρυθμής ε, ακόμα και τώρα δεν ρέουν τα κονδύλια. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας απασχολήσει, να δούμε πώς μπορούμε να εκταμιεύσουμε γρηγορότερα τα κονδύλια για τη γεωργία. Είναι σημαντικό να πάρουν οι άνθρωποι τα κονδύλια έτσι ώστε οι άνθρωποι να λάβουν αυτό το θετικό μήνυμα. Όχι να λένε μα δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς αφού δεν προκύπτει τίποτα το θετικό. Και κάτι άλλο. Μιλάμε συνεχώς για το ότι όλοι οι οικονομικοί ε, τομείς ε, πρέπει να επιτύχουν περισσότερα με λιγότερα μέσα. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε ε, το πώς μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα. Δηλαδή άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης που θα επιτρέπουν με τα λίγα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας να επιτυγχάνουμε περισσότερα. Ας πούμε τα κυλιόμενα ταμεία όπου εντωμεταξύ χρήματα σορεύονται και ανακυκλώνονται τα κονδύλια ε, για να μπορούν να έχουν καλύτερη χρήση. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε τέτοιου είδους ε, συστήματα, να έχουμε και καλύτερους ελέγχους. Τώρα δεν μιλάω για μικρές τράπεζες, αλλά για μεγαλύτερες τράπεζες. Με τις μεγαλύτερες τράπεζες μπορούμε να έχουμε ένα λογικό σύστημα ελέγχου για τη χρήση των κονδυλίων και για τα κριτήρια Έγκρισή του. σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πλουστευτούν οι διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία, να μην πρέπει κανείς να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά να αναθέτει και σε τρίτους ε, τον έλεγχο αυτό. Στη Γεωργία, ας πούμε, μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να πείσει κανείς ότι ορισμένες εργασίες μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους. Μπορούμε να θέσουμε ε, ορισμένες αρμοδιότητες σε τρίτους, υπεύθυνου τρίτους και δεν μπορούμε να μιλάμε για περιορισμό της ε, γραφειοκρατίας, αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα φοβούμαστε ότι θα χάσουμε τον έλεγχο. Αυτά και ευχαριστώ. Μάρτιν Όσλινγκ. Μάρτιν Όσλινγκ. Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής. Προηγουμένως ε, συζητήθηκε το θέμα της ε, συγχρηματοδότησης και πρέπει να το σκεφτούμε, να δούμε ε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε ορισμένα κράτη να εξαιρεθούν ακριβώς επειδή θα υπάρχει συγχρηματοδότηση. Κατανοώ ότι μερικοί εκμεταλλεύονται το θέμα της ε, συγχρηματοδότησης και δεν καταθέτουν προγράμματα επειδή δεν έχουν ε, όρεξη να το κάνουν αυτό. Ας πούμε η Γερμανία ε, δεν είναι φτωχή χώρα αλλά δεν προτείνεται η οικολογική καλλιέργεια στον δεύτερο πυλώνα και αυτό είναι πολιτική λόγη και όχι οικονομική. Γι' αυτό λοιπόν ορισμένα μέτρα στο δεύτερο πυλώνα πρέπει να είναι δεσμευτικά. Ε, πρέπει να υπάρχει εκτεταμένη οικολογική καλλιέργεια στον δεύτερο πυλώνα διότι ήδη ε, στον πρώτο πυλώνα διαπιστώσαμε ότι οι οικολογικές καλλιέργειες ε, καλύπτουν όλα τα κριτήρια της γεωργικής πολιτικής στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν η μία χώρα να προσφέρει κάτι τέτοιο και η άλλη όχι. Γενικά αυτό το κριτήριο του 25% πρέπει να εγγραφεί ως κριτήριο περιβάλλοντος δεύτερο πυλώνα. Και δεν είναι δυνατόν ε, ορισμένα κράτη να αποτελούν ε, υπόδειγμα ε, και άλλα πάλι να λένε εμείς δεν έχουμε χρήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δυστυχώς ε, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο δεσμευτικά και πρέπει να αλλάξει. Όσον αφορά το θέμα των μειονεκτουσών ε, περιοχών, συμφωνούμε, θα ξανασυζητήσουμε το θέμα όταν όλοι θα έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, κυρίως τα κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να δούμε κατά πόσον την, ε, θα δεχτούμε την πρόταση να δεχτούμε μόνο τους οκτώ παράγοντες. Πρέπει να υπάρχουν συνδυασμοί, γιατί αλλιώς θα υπάρξει μεγάλη, μεγάλη αναταραχή. Και η όλη ε, συζήτηση για τις μειονεκτούς περιοχές είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί σε πολλά κράτη. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε με κάποια δυνατότητα επιλογής στη μεταρρύθμιση. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, ε, στο δεύτερο πυλώνα αυτό είναι λάθος. Ε, δεν μπορεί να είναι μέτρο το οποίο χρηματοδοτεί από τον δεύτερο πυλώνα. Και πρέπει να διερωτηθούμε στη τελική ανάλυση ποιο επωφελείται. Μήπω οι ασφαλιστικέ εταιρείε επωφελούνται περισσότερο από τη γεωργία. Και επίση ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι με τι ασφάλειες... ο πενταετής ε, προγραμματισμός ε, είναι σχεδόν αδύνατος ε, για τα κράτη. Γιατί τι γίνεται αν προκύψει κάποιο ατύχημα και πρέπει να πληρωθούν αποζημιώσεις. Τότε δεν μπορούν πια να πληρωθούν, να χρηματοδοτηθούν άλλα προγράμματα. Νομίζω λοιπόν ότι οι ασφάλειες δεν ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα και εδώ συμφωνούν τα περισσότερα κόμματα. Και κάτι άλλο. Ε, νομίζω ότι εμείς ε, ως πολιτική ομάδα είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τον εισηγητή διότι ο δεύτερος πυλώνας ε, δεν είναι ουραγός του πρώτου αλλά είναι ο πυλώνας εκείνος με τον οποίο διαμορφώνουμε πολιτική και έχοντας μέτρα πρασινίσματος στον πρώτο πυλώνα αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιρούμε κάποια μέτρα από τον δεύτερο πυλώνα ισχύει το αντίθετο εμείς επιθυμούμε να ενισχύσουμε διπλά το πρασίνισμα, γι' αυτό πρέπει να μπει και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα και όχι το ένα εις βάρος του άλλου. Ευχαριστώ. Μισελ Νταντέν και μετά ο Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της συγχρηματοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης με την Κομισιόν κάθε χώρα να έχει την ελευθερία μέσα στα πλαίσια του συνολικού θεμά, θέματος των δίκτυ συγχρηματοδότησης, διότι πολλοί μπορούν να ζητήσουν υψηλότερη συγχρηματοδότηση με βάση τις εταιρικές σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν εδαφικά ή ακόμα και σε τομείς παραγωγής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κατευθυντήριο στοιχείο ως προς τις μειονεκτούσες περιοχές με βάση αυτά που είπε ο προλαλής σας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιμένουμε στα οκτώ βιοφυσικά κριτήρια που ισχύουν επί του παρόντος. Για παράδειγμα, στη χώρα μου Εάν την ε, περιοχή Σαμπάνι την θεωρήσουμε μειονεκτούσα περιοχή, θα ήθελα να μπορέσετε να το εξηγήσετε στη γαλλική κοινή γνώμη. Όπως είπε πολύ σωστά ο προλαλής σας, θα πρέπει να έχουμε σύμικτα κριτήρια έτσι ώστε να έχουμε έναν ρεαλιστικό χάρτη και να ανοιχνεύουμε τις βιωμένες δυσκολίες σε κάθε ε, εδαφική ενότητα ως προς τα ανώτατα όρια στις ορεινές περιοχές νομίζω ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι ύψης της σημασίας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι όμως το κουτί της Πανδώρας. Όλοι έχουμε συγκεκριμένες ιδέες και υπάρχει, έχουμε να κάνουμε με έναν μακρύ κατάλογο. Σε μία νύχτα αϊπνίας αποτίμησα την κατάσταση της χώρας μου. Έχουμε 980 εκατομμύρια ετησίως που δαπανώνονται και 290 ε, εκατομμύρια ε, δαπανώνται στις ορεινές περιοχές. και για τους νέους γεωργούς ε, χορηγούνται 280 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια για τη δασοκομεία και 350 που διατίθενται στις περιφέρειες που προωθούν τον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα και τις επενδύσεις στη γεωργία. Άρα τα έχουμε δαπανίσει όλα. Αν τώρα θα πρέπει να μπούμε στο ίδιο θέμα, στο ίδιο θέμα να εντάξουμε και την καινοτομία και τα ασφαλιστικά και το ασφαλιστικό και τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τα δάνεια θα πρέπει να επέμβουμε στην ΚΟΑ, στην κοινή οργάνωση της αγοράς και φοβάμαι ότι η μόνη γραμμή προσαρμογής αφορά τα αγροτικό περιβαλλοντικά. Εάν δεν έχουμε λοιπόν το πρασίνισμα στην, ε, στον πρώτο πυλώνα, δεν έχουμε το δικαίωμα να θυσιάσουμε τον αγροτικό περιβαλλοντικό ε, τομέα στο δεύτερο. Άρα επαναφέρουμε ε, πιστώσεις και δράσεις όπως τα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη δανειοδότηση στο πρώτο πυλώνα Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που κάνουμε με βάση τα δεδομένα των τεσσάρων εισηγητών, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικές θέσεις επί του θέματος. Σε σχέση με το θέμα που με απασχολεί, το μόνο δυναμικό στοιχείο είναι αυτά τα μία πιστοληπτικής ικανότητας για τις χώρες όπου μπορεί κανείς να συγχρηματοδοτεί σε περίοδο κρίσης. Εάν διαγράψουμε αυτό το μέσο, τότε χάνουμε τα μέσα που διαθέτουμε στην ΚΟΑ. Θα ήθελα τη γνωμοδότηση του εισηγητή γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεπείς όταν εργαζόμαστε επί του θέματος αυτού αλλά σας έδωσα τα δικά μας αριθμητικά στοιχεία. Αυτή, αυτό το προσθετικό εγχείρημα είναι ένα πραγματικό ζήτημα, δηλαδή προσθέτουμε και προσθέτουμε και προσθέτουμε, λέμε ότι θα πάει στον ένα ή στον άλλο πυλώνα, αλλά θα υπάρχει θέμα μέσων και για το τι μπορεί να επιτελέσει κάθε χώρα με βάση τον εθνικό προπολογισμό που θα πρέπει να πλαισιωθεί αν θέλουμε να υπάρχει μια συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε Μισελ, ο Σμιτ και ο κύριος Γιάζεβόλσκι στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, είμαι σκιώδης από την ομάδα μας και θα ήθελα να αρχίσω με ένα υπαρξιακό ζήτημα γιατί όταν μιλάμε για συγχρηματοδότηση μιλάμε για διαφορετική προσέγγιση ε, στην τελευταία μου θητεία ασχολήθηκα με τα περιφερειακά, την περιφερειακή ανάπτυξη και εδώ έχουμε μια διαφορετική ε, προσέγγιση. Πιστεύετε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένα υποβοηθητικό ε, μέσο της γεωργικής πολιτικής και ανάλογα με τα αν το δεχόσαστε ή όχι έχετε διαφορετική προσέγγιση ως προς την συγχρηματοδότηση σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κέστιγκερ για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ίσως θα μπορούσαμε να συνεδριάσουμε από κοινού με αυτή την Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο ε, μπορούμε να αποφανθούμε ως προς θέματα περιφερειακής ανάπτυξης πριν μιλήσουμε για συγχρηματοδότηση. Γιατί εντός Κοινοβουλίου υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και ας αφήσουμε τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν συντονίζουμε και αυτό το βλέπουμε σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία ε, προβαίνουν σε μία διάδραση και βλέπουμε ότι αυτοί οι οργανισμοί, ο, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες ορίζουν το πώς θα λειτουργήσει η ΚΑΠ και τα ανώτατα όρια με βάση την αγροτική ανάπτυξη και την περιφερειακή ανάπτυξη διότι θα υφίστανται πίεση οι προϋπολογισμοί μας και θα πρέπει να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτές τις συζητήσεις έτσι ώστε να είμαστε επικοδομητικοί. Θα επιλέξουμε ένα μικρότερο αριθμό βασικών τροπολογιών που θα συζητήσουμε με τον εισηγητή και θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτές. Δεν θα προβάλλουμε σωρία τροπολογιών γιατί θα πρέπει να ε, έχουμε δυνατότητα μόχλευση. Σε σχέση με τους ορισμούς του άρθρου 2, θεωρούμε ότι η καινοτομία και η αλυσίδα προμηθειών θα πρέπει να επεκταθεί ως προς τις συμβουλευτικές ε, υπηρεσίες. Θεωρούμε το άρθρο 16 θα πρέπει να αφορά και την αγροτική ανάπτυξη πέρα από την περιφερειακή και το ίδιο αφορά το άρθρο 17 για τα ποιοτικά σχέδια και το άρθρο 27 για τις οργανώσεις παραγωγών για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την αγροτική ανάπτυξη. Στο άρθρο 29 Μιλάμε για κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντικές. Θα θέλαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Το άρθρο 33 μιλά για τις ε, μειονεκτούσες περιοχές και έχουμε πολύ καλά παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν πολύ καλά και γίνανε βεβαίως και καταχρήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, αλλά να μην χάσουμε το σχετικό πλεονέκτημα σε ε, ευάλωτες περιοχές. Ως προς το άρθρο 34 για την ε, ευημερία των ζώων, την ευζοία, το έχουμε δείξει και σε άλλες εκθέσεις όπου υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας ως προς την ε, ευζοία, μεταφορά, υποδομές, σφαγή, σφαγές και ούτω καθεξής και τα άρθρα 42 και 44 αφορούν το πρόγραμμα Leader το οποίο χρησιμοποιήθηκε πολύ καλά και θα πρέπει να προσβλέπουμε σε αυτό έτσι ώστε αν δεν ε, απαλληφθεί τουλάχιστον ας μην το υπερδιορθώνουμε διότι αυτό δεν θα ήταν καθόλου αποτελεσματικό. Ευχαριστούμε Πασεβόλσκι και μετά Λουίς Άλβες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω αντιφατικές απόψεις σε σχέση με το δεύτερο πυλώνα, διότι δεν ξέρω κατά πόσο ο πρώτος πυλώνας και οι μοναδικές πληρωμές, οι ενιαίες πληρωμές δεν επιβαρύνουν το όλο σύστημα, αλλά βεβαίως οι αγρότες βασίζονται σε αυτές τις πληρωμές και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές υπάρχει μεγάλος φόρτος. Πολλές φορές δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Και πολλές φορές γίνονται μεγάλες ε, ουρές τους οργανισμούς ε, εκδήλωσης ενδιαφέροντος Έχουμε να κάνουμε με χίλιες εκμεταλλεύσεις στην Πολωνία, αλλά πολλοί άλλοι θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτό το πλαίσιο και δεν μπορούν. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με αυτά που είπε ο κύριος ε, Σμιτ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει επακριβώς ο δεύτερος πυλώνας εμπερικλείονται πολλοί στόχοι, υπερβολικά πολλοί και αυτό έχει μεγάλη σημασία να δούμε δηλαδή τι συμπεριλαμβάνουμε και τι όχι μέσα, στα βάσια μέσα με βάση τους στόχους που ορίζονται. Υπάρχουν ε, ορισμένες δραστηριότητες που έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν και γι' αυτό θα ήθελα στο δεύτερο πυλώνα να χρηματοδοτήσουμε τη γεωργία ε, κατά ορθολογικό τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ορίσουμε μία σειρά στόχων που να έχουν σχέση με τη γεωργία και όχι να μην έχουν άμεση σχέση. Μιλάμε για χρηματοδότηση σε περιφερειακές ε, ζώνες. Μιλάμε για επενδύσεις στην ευρυζωνική, στο ευρυζωνικό διαδίκτυο ή τουριστικές πληροφορίες στις αγροτικές περιοχές. Με αυτό αφορά την περιφερειακή πολιτική, όχι την αγροτική. Τι δουλειά έχει με την αγροτική. Πέρα από το γεγονός ότι ε, μιλάμε για συμμετοχή και αγροτικών περιφερειών. Δεν πρέπει να ε, ακολουθούμε μία σύμικτη πολιτική που να αναφέρεται και στην περιφερειακή και στην αγροτική μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ. Το ΚΑΠ ή ΚΑΠ αφορά χρήματα τα οποία θα πρέπει να έχουν ως τελικό παραλήπτη τους αγρότες. Το ίδιο αφορά και τις μικρές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν ΜΜΕ που λαμβάνουν πόρους από την ΚΑΠ και δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι δεν έχει σχέση με την ΚΑΠ θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν κατανοώ και την πρόταση αυτή που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της ΚΑΠ. Μιλάμε για τις μικρομεσαίες και μιλάμε για χρηματοδότηση των ΜΜΕ, αλλά από την άλλη πλευρά μιλάμε για χρηματοδότηση των αγροτών και των ε, κτηνοτρόφων που μεταφέρουν το ζωικό τους κεφάλαιο και που εξάγουν. Αυτό που θα πρέπει να προωθήσουμε είναι τις εξαγωγές μας Γι' αυτό οι στόχοι είναι αρκετά θολή και ασαφείς και θα ήθελα ο δεύτερος πυλώνας να χρηματοδοτείται και να αφορά χρηματοδοτήσεις που αφορούν αποκλειστικά την ΚΑΠ. Νέους αγρότες, μικρές εκμεταλλεύσεις, οικολογικές εκμεταλλεύσεις, αλλά καμία σχέση με την περιφερειακή πολιτική. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο γιατί και για την κοινή γνώμη είναι δύσκολο να συμμεριστεί αυτό το πλαίσιο. Φαίνεται ότι υπάρχουν υπερβολικά ποσά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αγροτική πολιτική. Γι' αυτό θα πρέπει να, να περιοριστούμε σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ. Θα ήθελα, λέει ο ομιλητής, ο κύριος Άλβες, να σταθώ σε δύο στοιχεία σε σχέση με την στρατηγική 2020 ε, και θα πρέπει να ε, δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ε, εναρμονισμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών. Μιλάμε δηλαδή για αγροτική δραστηριότητα κατά κύριο λόγο. Και στα πλαίσια του νέου πολιετούς πλαισίου θα πρέπει να μιλάμε για ένα στρατηγικό πλαίσιο που να συνάδει με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δηλαδή η διασταύρωση ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου, αλλά κυρίως περιφερειακού, διότι έχουμε να κάνουμε με πολιτικές και δράσεις εδαφικής χρειάς. Νομίζω λοιπόν ότι στις ε, εταιρικέ οικονομικές σχέσεις να μιλάμε για συμμετοχή των κρατών μελών και της Κομισιόν και να αναφερόμαστε σε περιφέρειες και αυτό έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε να ε, ε, υπερισχύει η αγροτική συνιστόσα και να μην ε, αποσπάται από τις προτεραιότητες. Ως προς τις μειονεκτούσες περιφέρειες, νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις περιφέρειες. και να μιλάμε για υποστήριξη η οποία να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και όχι εθελοντικό. Γιατί θα πρέπει να προβάλλουμε μία πιο συνεκτική εδαφική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Λουίς. Νομίζω ότι αυτό σχετίστηκε με την έκθεση Καρών στα πλαίσια της ε, περιφερειακής πολιτικής. Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πέντε σύντομες ε, παρατηρήσεις θέλω να κάνω όσον αφορά τα οικονομικά, ακόμα και αν δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορούμε να περάσουμε πάρα πολλά στον ε, πρώτο πυλώνα, αλλά και ο πρώτος πυλώνας κάποια στιγμή δεν χωράει τα πάντα, είναι και αυτός περιορισμένος. Το πρώτο πρόβλημα αφορά στη συγχρηματοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, υπενθυμίσω, ε, κάναμε μία πρόταση και είπαμε ότι τα μέτρα ε, που υπάρχουν στον πρώτο πυλώνα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αναφερόμαστε σε μέτρα περιβάλλοντος, σε επενδυτικά μέτρα ε, άρα δηλαδή δεν υπάρχει πλέον επιχείρημα να μην ισχύουν αυτά τα μέτρα. Και όσον αφορά στη χρηματοδότηση και στη συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου πρέπει να προσέξετε έτσι ώστε να μην υπάρξει τελικά ε, μεγαλύτερη ε, συμμετοχή του χρήστη. Δηλαδή στο τέλος ο Γεωργός ε, να πρέπει να πληρώνει περισσότερα χρήματα και αυτό να θεωρείται ε, ιδιωτικό κεφάλαιο. Ε, στο τέλος, όσον αφορά το facing out, κοιτάξτε, στο Ταμείο Συνοχής οι περιοχές οι οποίες φεύγουν από τις τους περιοχές την χάνουν ειδική χρηματοδότησης. Και θα ήθελα να δούμε κατά πόσο αυτό μπορούμε να το κάνουμε περισσότερο συμβατό αυτό το phasing out ε, για ε, πρώην μειονοτικές περιοχές ε, πρέπει να συμπεριληφθεί. Το τρίτο που θέλω να αναφέρω, αυτό νομίζω είναι έκκληση προς εμάς τους ίδιους. Δηλαδή να μην ξεχνάμε τον περιορισμό, τον της γραφειοκρατίας. Κατά τα άλλα, πρέπει να ξεκινήσουμε με θέματα γραφειοκρατίας και όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε διόγκωση της γραφειοκρατίας. Όσον αφορά τώρα το ΦΠΑ, δεν πρέπει να προαχθεί περαιτέρω. Για μένα λοιπόν το σημαντικό ερώτημα είναι ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα αφορά ε, την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν ξέρω ε, κατά πόσον αυτό αφορά τους ε, γεωργούς που δεν καταβάλουν ΦΠΑ. Όσον αφορά τις μειονεκτούσες περιοχές, Νομίζω ότι πρέπει ε, να το ξανασκεφτούμε το θέμα όλοι μαζί από κοινού, γιατί εδώ ασκείται ιδιαίτερα έντονη κριτική. Ε, είμαστε όλοι ανικανοποίητοι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτό το θέμα των μειονεκτουσών περιοχών να το εξαιρέσουμε με την έννοια ότι πρέπει να έχουμε χρόνο να σκεφτούμε το όλο θέμα. Γιατί πιστεύω ότι δεν εξυπηρετούμε τις μειονεκτούσες περιοχές να συζητάμε όλο αυτό το τεράστιο πακέτο. Ίσως δεν είναι το καλύτερο αυτές να τις αφαιρέσουμε και να τις συζητήσουμε κάπου ξεχωριστά όταν θα μιλήσουμε για την αγροτική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξεκινάω λοιπόν ε, από κάτι που ε, υπήρξε εδώ, το θυμάμαι ότι υπήρξε εδώ, όταν ξεκίνησε η θητεία μου. Όταν ελέγχθη ότι θα πρέπει να φέρουμε κάποιον επιτόπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φέρνουμε κάποιον στα σημεία της καταστροφής. Αναφέρομαι λοιπόν, καταλάβατε, σε εγκαταλελειμμένες περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης ε, προσοχής. Αναφέρομαι στις ε, διάφορες τοποθεσίες ε, που μπορεί κανείς να βρει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το πρασίνισμα δεν πρέπει να είναι κάτι το γενικευμένο, αλλά πρέπει να είναι μια πρόταση πρασινίσματος. Κυρίως στις γεωργικές περιοχές τις εγκαταλελειμμένες και μειονεκτούσες γεωργικές περιοχές, εκεί θα μπορούσε κανείς να επιτύχει περισσότερα με εξειδικευμένα μέτρα για να επιτύχει μια νέα επιχειρηματικότητα. Ένα μείγμα δραστηριοτήτων που δεν θα είναι μόνο γεωργικές, αλλά και άλλες. Και Ίσως ε, με τον τρόπο αυτό ε, μπορεί κανείς ε, να φέρει κάποια ισορροπία. Ίσως θα μπορούσαμε να φέρουμε και από τις πόλεις ανθρώπους ε, προς ε, τις ε, μειονεκτούς περιοχές και στην Ήπεθρο. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι ίσως μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν την διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις μεγάλες εκτάσεις με λίγους ανθρώπους και αυτό είναι μια πραγματικότητα όπου ο καθένας θα μπορούσε να κάνει τη δική του την επιλογή. Ευχαριστούμε. Θα κλείσει ο κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με κάποιους ε, από τους προλαλήσαντες και θα ήθελα μάλιστα να προσθέσω κάποιες παρατηρήσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, πιστεύω ότι η ενίσχυση για μη γεωργικές δραστηριότητες, και αναφέρομαι στο άρθρο 20, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει την συμμετοχή μικρών και μεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων, αλλά δεν θα έπρεπε να περιορίζει και την συμμετοχή των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων ο περιορισμός των επενδύσεων της στήριξης ε, σε διαρθρωτικά προβλήματα δεν είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Θα έπρεπε η υποστήριξη αυτή να ε, δίδεται σε όλους τους γεωργούς, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα στην Ευρώπη, στην παγκόσμια αγορά. Κάτι ακόμη το οποίο αναφέρθηκε ήδη σήμερα η χρήση των ε, επενδυτικών κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα και ότι δεν έχει πολύ σχέση αυτό με τη γεωργία. Νομίζω ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να διαγραφούν. Αναφέρομαι στην ε, διαδικασία ε, μη ε, γεωργικής παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα 1 της συνθήκης. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει αυτό μόνο για τα βιοκαύσιμα και για την ε, βιολογική ενέργεια. Έτσι θα έπρεπε να έχουν τα πράγματα. Επίσης πιστεύω ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ε, τις ε, περιοχές ε, υπομετάβαση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Περιοχές δηλαδή που πρώτη φορά περνούν το 75% του μέσου ΑΕΠ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία λοιπόν. Τώρα θα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Και μετά ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και τα σχόλια που ακούστηκαν. Ορισμένα ζητήματα είναι κατά καθαρά πολιτικού χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλει να αρκεστεί σε ε, σχόλια τεχνικού χαρακτήρα περισσότερο και να εξηγήσει κάποια στοιχεία της πρότασης. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω με τις ε, ε μειονεκτούσες περιοχές που έχουν φυσικούς περιορισμούς υπήρχαν κάποια ερωτήματα σε σχέση με την ε, πρόοδο της οριοθέτησης ε, του ορισμού αυτών των ε, περιφερειών. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη επεξεργάζονται τον χαρακτηρισμό των ε, περιοχών αυτών ε, με ε, συγκεκριμένους όρους, όπως για παράδειγμα περιφέρειες στις οποίες υπάρχουν φυσικοί περιορισμοί και μάλιστα μέσω λεπτομερών χαρτών. Έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη τα στοιχεία αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι εντελώς προκαταρκτικά για την ώρα αυτά τα έγγραφα. Τα κράτη-μέλη σε γενικές γραμμές είναι διστακτικά ε, ως προς τη δημοσίευση των ε, εγγράφων αυτών. Κάποια κράτη-μέλη όμως τα δημοσιεύουν, ε, τέλος πάντων ε, σε περιορισμένο βαθμό, σε κάποιους ευρωβουλευτές για παράδειγμα. Οπότε, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να οργανώσει ένα ε, μια συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο ε, Ευρωβουλευτή ώστε να μπορεί να γνωρίζει ε, το κοινοβούλιο καλύτερα τι συμβαίνει. Βέβαια ο χαρακτηρισμός των περιοχών αυτών δεν είναι οριστικός. Ακόμη είναι υπό επεξεργασία γιατί κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζεται λοιπόν η εργασία επί του θέματος αυτού, όμως μπορούμε ήδη να διαθέσουμε κάποιες πληροφορίες που έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας. Η προσπάθεια αυτή καλύπτει και μια προσπάθεια από πλευράς κρατών μελών να ε, αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα που ήδη αναφέρθηκε, ε, το πρόβλημα της περιοχής ε, που αναφέρθηκε, δηλαδή τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, εξαιρέσουν μια περιοχή ε, που δεν είναι μειονεκτούσα περιοχή από μια ευρύτερη περιφέρεια ε, που θεωρείται γενικά μειονεκτούσα. Μπορούμε λοιπόν να οργανώσουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών με τους ευρωβουλευτές για το θέμα αυτό. Κάτι ακόμη για την ανακατανομή των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα. Για αυτό το θέμα μόνο να επιβεβαιώσω μπορώ ότι δεν θα υπάρξει πρόταση από πλευρά Επιτροπής για την ανακατανομή ε, του προϋπολογισμού από το δεύτερο πυλώνα, το δεύτερο πυλώνα για το 2014 ως το 2024. Η, η κατανομή θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με τους στόχους πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατανομή. Οπότε, πιστεύω ότι αυτές είναι οι αποσαφηνίσεις που χρειάζονται για την ώρα σε σχέση με ε, τις διατάξεις Τώρα το ζήτημα του 25% ε, της ε, ε, του επίπεδου της χρήσης ύδατος για προγράμματα άρδευσης. Είναι βεβαίως προφανές ότι μέλλον, ε, στο μέλλον θα έχουμε όλο και λιγότερους πόρους και πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ε, αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς τον κανονισμό προτείνουμε νέες επενδύσεις ε, για την άρδευση, 25% εξοικονόμηση δηλαδή στη χρήση ύδατος σε σχέση με το πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 25% της μείωσης της χρήσης των υδάτων ε, ε, ήδη υφίσταται στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης και των σχετικών κανόνων. Υπάρχει δηλαδή ε, μία εξαίρεση στον κανονισμό που επιζητά μείωση κατά 25% της χρήσης του νερού για αρδευτικά προγράμματα. Για προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς προπολογισμού. Ένα ακόμη ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση του κινδύνου και το λόγο για τον οποίο τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου βρίσκονται στο δεύτερο και όχι στον πρώτο πυλώνα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα της διαχείρισης κινδύνου έχουν πολυετή χαρακτήρα και γι' αυτό προτείνεται η χρήση κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα, πολυετή προγράμματα δηλαδή για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού και όχι να ε, εστιαστούμε μόνο στον πρώτο πυλώνα. Αυτό στο πλαίσιο του άρθρου 68. Υπάρχει θετική αξιολόγηση επίσης του προγράμματος Leader. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Leader, επί τη βάση της ε, πρότασης αυτής, θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης το προγράμματος Leader από ε, άλλες ε, πηγές, όπως για παράδειγμα μέσω των ομάδων τοπικής δράσης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ευελιξίας ε, του προγράμματος Leader. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι συμφωνούμε σχεδόν όλοι ότι μεγαλύτερο συντονισμός ε, χρειάζεται μεταξύ των ε, πηγών χρηματοδότησης και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικές οι δημόσιες συμβάσεις ε, για την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφερθεί επίσης το ότι πολλές λεπτομερείς, ε, λεπτομερή ε, θέματα που αναφέρθηκαν σήμερα έχουν λυθεί σε επίπεδο προγραμματικής περίοδου όταν τα κράτη-μέλη θα προετοιμάσουν τα προγράμματά τους. Οπότε μπορούν να, ασχοληθούν και με το ζήτημα της στρατηγικής. Για παράδειγμα, καινοτομία. Υπόθηκε ότι η καινοτομία ε, θα, θα προέρχεται μόνο από το κάπινγκ, δηλαδή από τις οροφές. Αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα, ένα βασικό τμήμα του αναπτυξιακού μας προγράμματος και βεβαίως τα κράτη-μέλη θα ήταν ευπρόσδεκτα αν ε, αντιμετώπιζαν το πρόβλημα αυτό και στα δικά τους ε, εθνικά προγράμματα, στη δική τους εθνική στρατηγική. Αν χρησιμοποιηθούν δηλαδή πόροι για την καινοτομία στο πλαίσιο ε, συνεργασίας για την καινοτομία. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για, την... για τα προγράμματα αυτά. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τον συνάδελφό μου να συμπληρώσει τα δικά μου λεγόμενα. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπληρώσω. Σχεδόν όλα τα είπατε. Θα ήθελα απλώς να τονίσω το γεγονός ότι όσον αφορά την καινοτομία είναι ένα πάρα πολύ ειδικό θέμα 100% προέρχεται από το κάπινγκ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν υπάρχουν για την καινοτομία. Για όλα τα μέτρα, για όλες τις προτεραιότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση αυτή, ενισχύεται από τα κονδύλια του κάπινγκ. Αυτά ε, αποτελούν το 100%, τα υπόλοιπα Και όπως ε, είπατε και εσείς ε, κύριε Γενική Διευθυντή, ε, στο πλαίσιο του προγραμματισμού το κράτος μέλος πρέπει να κάνει μία ανάλυση και πρέπει να ορίσει τη στρατηγική του και θα επιλέξει τα μέτρα που ε, ε, εκπληρώνουν τις ε, συγκεκριμένες ποσοτικοποιημένες προτεραιότητες. Κύριε Ντοντέν, λοιπόν, δεν θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι τα, χρώματα θα, τα χρήματα θα διατεθούν για τα 20 μέτρα. Όχι, τα χρήματα θα διατεθούν για τα μέτρα που θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στις επιλεγμένες προτεραιότητες. Σήμερα είναι 20, το 2007 με 2013 ε, ήταν 40. Όσον αφορά τώρα το θέμα του χρηματοδοτικού μηχανισμού, ναι, είναι γεγονός ότι και εκείνη υπησέρχεται για να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουμε και όταν, μιλάω, ε, όταν λέω έχουμε, μιλάω για τα κράτη-μέλη. Από εθνικής πλευράς τώρα, νομίζω ότι τα μέτρα αυτά που προανέφερα μπορούν να βοηθήσουν. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Α! Το άρθρο 18 και το άρθρο 20. Ναι. Εκεί υπάρχει μία στόχευση. Μία στόχευση αλλά μόνο για τις εκμεταλλεύσεις που έχουν προβλήματα αναδιάρθρωσης και εκεί αναφέρονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει ε, περιορισμός. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε λοιπόν τους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον εισηγητή, στον Λουίς, για να κλείσει το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Είπαμε πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους που πήλαν το λόγο για τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά τους. Θα ληφθούν υπόψη. Να ευχαριστήσω επίσης ε, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχόλιά τους και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να αποδεχθεί και τις δικές μας παρατηρήσεις ε, για τον εμπλουτισμό της συζήτηση. Ξέχασα να σας πω το ευαίσθητο θέμα θα είναι η κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των κρατών μελών είπε ότι όλα τα κράτη-μέλη που πρέπει να συνεισφέρουν ε, στην ε, εξισορρόπηση του πρώτου πυλώνα δεν θα έπρεπε να ε, τιμωρηθούν στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Οπότε πρέπει να υπάρξει, να οριστεί μια βασική αρχή που θα εξασφαλίσει ότι κανένας δεν θα τιμωρείται ουσιαστικά δεδομένου ότι είναι ένα ζήτημα πολύ ευαίσθητο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ισχύσει η αρχή της αλληλεγγύης και ε, ώστε η, αλληλεγγύη να μην τεθεί ένα αμφιβόλο. Πολύ ωραία, μπορούμε τώρα να περάσουμε στα άλλα θέματα της σημερινής διάταξης. Τα σημεία 6 και 7 ε, θα τα αναβάλουμε γιατί η συγγήτρια δυστυχώς ε, έχει εμπλακεί και δεν μπορεί να φύγει από την ε, Επιτροπή των Γυναικών. Αλλά έτσι και δεν υπάρχουν και πάρα πολλά νέα από την τριμερή συζήτηση. Περιμένουμε την Προεδρία της Δανίας για να δούμε αν μπορεί να μας ε, πει κάτι. Εν πάση περιπτώσει αναβάλλεται αυτό το θέμα στην ε, επόμενη συνεδρίαση. Ε, θα δώσουμε τότε το λόγο για να μας ενημερώσει η Τελευταίο σημείο το οποίο παραμένει σήμερα, το σημείο υπαριθμών 8, είναι ένα κείμενο προσαρμογής με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εισηγητής ο κύριος Τζανκάρλος Σκοτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Η πρόταση λοιπόν αφορά ε, αυτό το ε, δίκτυο λογιστικής ε, πληροφόρησης που συστήθηκε για να καλύπτει την ε, γεωργία, κυρίως όσον αφορά την, ε, τα εισοδήματα και την ανάλυση ε, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό λοιπόν το σύστημα εξελίχθηκε και επεκτάθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα εναρμονισμένο αρχείο το οποίο προσφέρει μικροοικονομικά στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη το σύστημα αυτό το λογιστικό που λέγεται ρίκα σε συντομογραφία αξιολογεί τις γεωρικές πολιτικές με την έννοια ότι ε, συγκεντρώνει στοιχεία για τα εισοδήματα και γενικότερα για τις γεωρικές εκμεταλλεύσεις. Αυτή τη στιγμή το δείγμα περιλαμβάνει 80.000 από τα 6 εκατομμύρια γεωρικές εκμεταλλεύσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή το σύστημα αυτό επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει την οικονομική ε, πολιτική πολιτική ε, και να υπολογίσει κάποιους δείκτες ε, που έχουν σχέση με το εισόδημα, την παραγωγικότητα και το κόστος ε, παραγωγής. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις της καινής γεωργικής πολιτικής. Αυτά τα δεδομένα στηρίζονται και από άλλα Ινστιτούτα έρευνας που ασχολούνται με τη γεωργία. Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού δεν αγγίζει ουσιαστικά αυτό το σύστημα της λογιστικής και ο στόχος ε, είναι να ευθυμεγραμμιστούν ε, οι διαρμοδιότητες της Επιτροπής με το 290 και 291 σχετικά με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Οι βασικές αλλαγές είναι η κατάργηση του παραρτήματος 1 που περιλαμβάνει τον κατάλογο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυτό ε, για να υπάρξει απλούστευση από τη στιγμή που ο ίδιος κατάλογος υπάρχει ήδη στον κανονισμό 1291. Ε, η Κομισιόν προτείνει στο μέλλον να υπάρξει ε, προσαρμογή τα κράτη-μέλη επίσης δεν θα είναι υποχρεωμένα να στέλνουν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ένα κατάλογο ε, το τρίτο είναι κατάργηση του πλαφών αναφέρομαι στο άρθρο 5 του κανονισμού που λέει ότι θα πρέπει στο σύστημα ε, αυτό να συμμετέχουν ε, κατά το ανώτατο όριο 5.000 εκμεταλλεύσεις. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός και το σύστημα παραμένουν ανοιχτά προς όλους. Εξάλλου οι ε, αρμόδιες αρχές και η συνεργασία με τα ε, λογιστικά γραφεία και με το σύστημα θα πρέπει αυτό να είναι ενιαίο σε όλα τα κράτη με λοιπά και το σχετικό άρθρο. Η νέα λοιπόν πρόταση προτείνει να παραγραφεί όμως αυτή η παράγραφος γιατί είναι απαρχαιωμένη. Σε γενικές λοιπόν γραμμές εγώ στηρίζω αυτές τις αλλαγές και η μόνη ε, με, τροπολογία που προτείνω είναι να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ιστότοπος ε, που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτού του συστήματος. Σας ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω αν επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο. Αν δεν υπάρχουν ε, παρεμβάσεις και αν δεν θέλει να παρέμβει και η Επιτροπή, πάρα πολύ ωραία. Α, μισό λεπτό. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπέβαλε την πρόταση αυτή. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο εισηγητής, με τα περισσότερα. Απλώς θα ήθελα να πω το εξής, ότι υπάρχει ένας ιστότοπος ε, για το θέμα αυτό της λογιστικής πληροφόρησης ε, που είναι διαθέσιμος σε όλους, στο κοινό, στο κράτη-μέλη και μάλιστα υπάρχει και στον ιστότοπο, στο, στον ιστότοπο Ευρώπα. Ευχαριστώ. Uh, Mr. Ok, chiedo scusa ma c'ho il commissario che mi sta aggiornando su una questione abbastanza delicata. Ενημερώθηκα για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε για σήμερα. Επόμενη συνεδρίαση στις 23 Απριλίου και στις 24 Απριλίου από τις 9 και τα απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.